Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινούμε. Έχουμε ακόμη να ε, εξετάσουμε διάφορα θέματα και ε, υπάρχει το θέμα των υποδομών για το 2020 το οποίο ξεκινήσαμε χθες αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον συγητή κύριο Σούζα για να μας κάνει την εισαγωγή στο θέμα. Και... Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι η έκθεση αυτή ήταν σημαντικό όταν αποφασίσαμε να το εκπονήσουμε, αλλά με την καταστροφή τώρα στην Ιαπωνία, τα ζητήματα αυτά είναι ακόμη πιο επίκαιρα. Αυτή τη στιγμή η αντίδραση της Ευρώπης ε, σε αυτή την καταστροφή στην Ιαπωνία πρέπει να είναι σαφής. Είδατε την έκθεση αυτή σε όλες τις γλώσσες. Αλλά η έκθεση δεν επιλύει τα προβλήματα, όλα τα ενεργειακά προβλήματα που υφίστανται. Αναλύει κάποια από αυτά, αλλά δεν είναι δυνατόν να τα αναλύσει όλα διεξοδικά. Εμείς θελήσαμε να ορίσουμε τι ακριβώς εννοούμε ενεργειακή υποδομή. Αυτό ήταν ο στόχος της εν λόγω έκθεσης. Δεν πρόκειται Δεν αφαιρθούμε σε, όλα, σε όλους τους όρους ε, που αφορούν την ενέργεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε ό,τι αφορά την ε, δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού δικτύου. Οπότε, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, ότι στο ενεργειακό επίπεδο τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η νομοθεσία, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σεβαστούμε και τις συνθήκες. Αυτή είναι η έκθεση. Αυτό είναι το νόημα της έκθεσης και θα προσπαθήσω να σας πω σε τι ακριβώς επικεντρώνεται. Πρέπει να αναπτύξουμε τις ενεργειακές υποδομές, ε, πρέπει να αποφύγουμε εθνικό κατακαιρματισμό, πρέπει να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρέπει να προωθήσουμε την αποτελεσματικότητα των ενεργειακών πηγών, να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό μας σε ενέργεια, όπως επίσης και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα κράτη-μέλη, που ε, εξαρτώνται από έναν μόνο ενεργειακό προμηθευτή. Η ιδέα μία δικτύωσης ε, των διαφόρων ενεργειακών υποδομών που συνδέουν τα διάφορα κράτη-μέλη είναι απαραίτητη αν θέλουμε να υπάρχει πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, που είναι επίσης ένας στόχος της συνθήκης. <coughs> Σύμφωνα με την έκθεση, πρέπει να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε επίπεδο. Έχουμε όμως την τάση να πιστεύουμε ότι υπάρχουν κανόνες στην Ευρώπη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεπώς όλοι οι κανόνες που υπάρχουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρομαι κυρίως στο τρίτο ενεργειακό πακέτο αλλά και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες που υπάρχουν για το θέμα της ενέργειας πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν. Είναι επίσης σημαντικό και το αναφέρει και το κείμενό μου, Πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ των στόχων της ενεργειακής πολιτικής ε, και της ε, πολιτικής για το κλίμα. Και όλα αυτά να συνάδουν με τα ε, μέτρα και τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν σε διάφορους τομείς οι σχετικές πολιτικές, οι σχετικές με την ενέργεια πολιτικές, να έχουν μια, ένα, συνεκτικό, ένα συνεκτικό στόχο. Πολύ σημαντικό είναι και το θέμα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Είμαστε πάρα πολύ εξαρτημένοι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο από ξένους προμηθευτές. Επομένως, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και επίσης υπάρχει επίσης και η κατεύθυνση της η ε, ε, προσανατολισμός ε, των απαιτήσεων των ενεργειακών των πολιτών και αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερως σε όλες τις ενεργειακές επενδύσεις που κάνουμε. Τι, τι, τι απαιτήσει υπάρχουν σε ενέργεια και πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε με την εξοικονόμηση ενέργειας. Και γι' αυτό είναι επίση σημαντικό να ξέρουμε ακόμη καλύτερα τις υποδομές που έχουμε στη διάθεσή μας. Και αυτό με οδηγεί στο επόμενο σημείο που αναφέρω στο κείμενό μου, και αυτό είναι η ανάπτυξη των ευφυών δικτύων. Εχθές είχαμε μάλιστα και μία δημόσια ακρόαση με εμπειρογνώμονες. το σχέδιο έκθεσής μου. Συμπεριλαμβάνει κάποια, κάποιες από τις ιδέες που ακούστηκαν και από τους προσκεκλημένους μας εχθές. Η ανάπτυξη αυτών ε, των ε, ενεργειακών ε, δικτύων, των ευφυών δικτύων, σημαίνει ευφυής πόλης. Συχνά ξεχνούμε ότι η ενεργειακή πολιτική συμπεριλαμβάνει πολλούς εταίρους. Την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό ακριβώς έχουμε αναλάβει το θέμα αυτό. Και τα κράτη και οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και η Ευρωπαϊκή Δήμη είναι εταίροι στην προσπάθεια αυτή. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ενεργειακή πολιτική χωρίς να υπάρχει ευαισθητοποίηση από πλευράς δημάρχων των κατοίκων των πόλεων. Εκείνοι είναι υπεύθυνοι προκειμένου να ζητήσουν την εξοικονόμηση ενέργειας και να προσπαθήσουν να την επιτύχουν. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με τις προσπάθειες που κάνει κάθε πόλη σε ζητήματα μεταφορών, για παράδειγμα. Επομένως, ευφυείς μεταφορές και ευφυείς πόλεις. Χρειαζόμαστε συνεπώς να μπορούμε να βασιζόμαστε στις τοπικές αρχές. Και όλα αυτά βέβαια συνδέονται και με την ιδέα μιας αποκεντρωμένης διαχείρισης των ενεργειακών υποδομών. Στο παρελθόν όλα ήταν αποκεντρωμένα σε σχέση με την ενέργεια. Και σήμερα, εκτός από την αναπόφευκτη αυτή αποκέντρωση για την παραγωγή ενέργειας, που είναι και αυτή σημαντική, χρειαζόμαστε μία ακόμη πιο αποκεντρωμένη προσέγγιση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι ο καταναλωτής είναι παράγον πολύ βασικός όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα. Και αυτό βέβαια συνδέεται και με αυτό που μόλις σας είπα. Δηλαδή ότι οι ευφυείς πόλεις θα δώσουν τη δυνατότητα μίας πολιτικής ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας. Από το 1985 αναφέρουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να τονίζουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία. Δεν χρειάζεται να σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες, ούτε να αναφερθώ σε όλα όσα έχω συμπεριλάβει στο κείμενό μου. Άλλωστε στο κείμενο είναι όλα πολύ σαφή. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι διάφορες πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλυφθούν σε σχέση με όλα αυτά τα σημεία που αναφέρω στην έκθεσή μου. Και οι προτάσεις σας είναι ενδιαφέρουσες και ευπρόσδεκτες. Μιλήσαμε για τον εφοδιασμό, για τους κλιματικούς στόχους, ε, η προσφυγή σε αποδεδειγμένες τεχνολογίες. είναι θέματα τόσο σημαντικά που ποτέ δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία και τις αδειοδοτήσεις. Εκτές ακούσαμε δύο εμπειρογνώμονες σε σχέση με το θέμα αυτό. και χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα όλα όσα είπαν. Άλλωστε έχω συμπεριλάβει το στοιχείο αυτό στην έκθεσή μου. Πρέπει οπωσδήποτε να διευκολύνουμε τη διαδικασία. για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε και την άμεση εφαρμογή αυτών των διαδικασιών, προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε και την πρόσβαση στις δημόσιες, στις δημόσιες διοικήσεις. Μιλάμε επίση και για τη συμμετοχή του πολίτη. Και από την αρχή κάθε προγράμματος είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας υποστηρίζουν οι πολίτες και πρέπει να ζητήσουμε την υποστήριξη αυτή από την αρχή. Όταν ένα πρόγραμμα δεν είναι <coughs> όριμο ακόμα, και όταν ακόμη υπάρχουν ανοιχτές όλες οι δυνατότητες. Έτσι έχουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά πώς πάνε τα πράγματα όταν δεν υπάρχει υποστήριξη των πολιτών. Πρέπει να εξηγούμε λοιπόν στους πολίτες ότι οι συνέπειε που θα υποστούν δεν είναι τεράστιε λόγω της εφαρμογής ενός προγράμματος. Εχθέ στην ακρόασή μα. οι εμπειρογνώμονε ανέφεραν ιδέες ε, οι οποίες περιλαμβάνονται και στο σχέδιο έκθεσης, όπως για παράδειγμα ότι η αγορά είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να ε, συλλάβουμε τα προγράμματα αυτά και να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε. Επίσης, είναι σημαντικό να έχουμε και μία πολιτική τιμολογιακή διαφανή. Πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για τη χρηματοδότηση. οι επιχειρήσεις δεν ζητούν τόσο, δεν είναι τόσο απαιτητικέ σε δημόσια κονδύλια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και ποιες θα είναι οι ρυθμίσεις για το μέλλον. Πρέπει να ξέρουμε τι δημόσιες δαπάνες μπορούν να υπάρξουν όταν υπάρχει ένα ε, κοινό όφελος και αυτό είναι ένα τρόπος για να προσελκύσουμε δημόσιες επενδύσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν, πρόκειται για μία έκθεση που είναι πάρα πολύ σημαντική Αλλά μετά τις ε, αποκαλύψεις ε, που ακούσαμε χθες, μας είπε και η Επίτροπος ότι είναι ακόμη πιο σημαντικές ε, αυτές οι πολιτικές. Χρειάζεται οπωσδήποτε η δικτύωση ενεργειακή για να έχουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Και ο στόχος αυτός είναι ένας στόχος αναπόφευκτος. Εμείς εδώ είμαστε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Πρέπει να διαλέξουμε το δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Και είναι πραγματικά μια πρόκληση για μας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για τις προτάσεις τους Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που δεν ήταν συνεισηγητέ, αλλά πραγματικά μου υπέβολαν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσε παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα έχουμε ήδη 13 συναδέλφους που ζητούν ε, το λόγο και μέχρι τις 10 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση άρα έχουμε δύο λεπτά για κάθε ομιλητή διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε δίνω πρώτα ε, το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές και πρώτα είναι ο Κάρενς. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Ευχαριστώ τον εισηγητή. Είναι καλό που έχουμε τη συζήτηση αυτή τώρα και φαντάζομαι ότι αυτές οι τροπολογίες δεν θα αλλάξουν ούτως ή άλλως την ουσία της έκθεσης αλλά θέλουν να διευκρινίσουν ορισμένα θέματα και ένα από αυτά τα οποία θα ήθελα να τονίσω γιατί το σημείωσα εχθές στη δημόσια ακρόαση που παρακολουθήσαμε ήταν ότι κανείς σχεδόν δεν μιλούσε για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό που είναι η κοινή αγορά που θα έπρεπε ουσιαστικά να είναι ο στόχος για τον οποίο η Ευρώπη θέλει να δημιουργήσει ένα κοινό δίκτυο για να επιτύχει μια τέτοια κοινή αγορά και να αυξήσει τον ανταγωνισμό υπέρ των καταναλωτών, να έχει ένα σταθερό πλαίσιο και τη δυνατότητα ε, για τις ιδιωτικές εταιρείες να επενδύσουν στην υποδομή. Οπότε ορισμένες από τις τροπολογίες ε, στις οποίες θα υποβάλλω ε, θα ασχοληθούν με τα θέματα αυτά. Όχι ότι δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο αλλά πρέπει να είναι ίσως στο επίκεντρο και όταν ε, το, η Επιτροπή θα φέρει στο Κοινοβούλιο την νομοθετική ε, πράξη να γνωρίζει ότι αυτός είναι ένας σαφός, σαφής στόχος για αυτό το θέμα. Δεν θέλω να περάσω τα δύο λεπτά, οπότε μετά τα δύο μου λεπτά, όταν θα επισέλθουμε στις λεπτομέρειες, θα επανέλθω. Ευχαριστώ. Η κυρία Ριέρα Μαντουρέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, για άλλη μια φορά ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σόζα Βάγνερ για την δουλειά του και για την διεξοδική του παρέμβαση. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τις προτάσεις του και θα συμφωνήσω και με τα σχόλια που έκανε στην παρουσίασή του. Δηλαδή θεωρώ και εγώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα αυτό δεδομένων μάλιστα και των ε, συνθήκων που κυριαρχούν σήμερα. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης θέλω να κάνω ορισμένα σχόλια. Και να αναφερθώ και στις τροποποιήσεις που έχει προτείνει η ομάδα μου. Κανείς δεν θα παραξενευτεί με την υποβολή τροπολογιών που που έχουν να κάνουν με το 10% για τις δυνατότητες ε, διασύνδεσης. Μας ενδιαφέρει να επιδιώξουμε τον ε, στόχο αυτό σε σχέση και με τους στόχους ε, της στρατηγικής του 2020 για την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές και την ε, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ βλέπουμε ότι στο ευρωπαϊκό δίκτυο πρέπει να συνεχιστούν σοβαρές επενδύσεις στο σύστημα υποδομών μας Και ήδη από τους προσκεκλημένους μας θες μια επιβεβαίωση για όλα αυτά και για την ανάγκη μιας ευρωπαϊκότερης θεώρησης του όλου θέματος. Χρειάζεται ένα έγγραφο στρατηγικό από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταφέρουμε πραγματικά να επιτύχουμε αυτό το στόχο του 10%. Ήθελα επίσης να πω ότι στηρίζουμε την πρόταση του εισηγητή να εξεύρουμε μηχανισμούς χρηματοδότησης που να βασίζονται στην αγορά. Δεν αρκεί όμως να έχουμε ομόλογα για να χρηματοδοτηθούν από αυτά κάποια προγράμματα, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει ακριβώς και με τα καύσιμα. Σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στηρίζουμε την ε, πρόταση του συγητή και Πρέπει επίση να έχουμε κατά νου ότι εδώ υπάρχει και ένα ευρύτερο στόχο με τον ε, μακρύτερο ορίζοντα του 2050. Θα εκφράσω επίσης τη στήριξή μου για τα πιλωτικά σχέδια που αφορούν το νότο της Ευρώπης και επίσης ως και όδηση εισηγήτρια να επισημάνω ότι είναι πραγματικά ιδιαίτερα επικοδομητική και θετική η στάση του εισηγητή. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Θα καταλήξουμε πιστεύω σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, να συγχαρώ τον κύριο Σόζα Βάγκνερ για την διεξοδική και εξαιρετική του έκθεση. Θέλω να πω ότι στηρίζω πλήρω τις προτάσει του. Λίγα σχόλια απλώ. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλούμε για τι επενδύσει τι υποδομές και τον σχετικό προγραμματισμό, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα το μακρύτερο ορίζοντα του 2050. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον οδικό χάρτη για το 2050, υπέβαλε κάποιε προτάσει. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει συνοχή και συνέπεια μεταξύ όλων μας των στόχων και μεταξύ της στρατηγικής του 2050 ε, με την θεώρηση για το του 2020 με την θεώρηση για το 2050 και με τους υπόλοιπους στόχους μας για τον περιορισμό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, για την ενεργειακή ασφάλεια και την ε, ενεργειακή προμήθεια, για την ε, χρηματοδότηση τώρα η φιλοσοφία μας παραμένει ότι θα πρέπει να είναι η αγορά ε, αυτή που θα καθορίζει την ε, κατεύθυνση των επενδύσεων. Και αυτό για να μπορεί να δικαιολογηθεί και η κρατική βοήθεια. Επίσης για τα ευρωπαϊκά ομόλογα βλέπουμε αυτό να είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λύση και πιστεύουμε ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να το σκεφτεί αυτό προσεκτικά. Θα μπορούσε να γίνει ένα καθοριστικό δημοσιονομικό εργαλείο για να εξεύρουμε αυτά τα κονδύλια που θέλουμε τόσο πολύ να επενδύσουμε. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα της ιδιοκτησίας των υποδομών ενέργειας, οι εταιρείε ή οι θυγατρικες τους, η διαχείριση των εταιριών αυτών. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι διαφανή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να έχουμε τις επαρκείς νομικές ε, εγγύησεις για να είμαστε διασφαλισμένοι εδώ και να ξέρουμε και ποιος έχει πρόσβαση σε κρατική επιχορήγηση. Επίσης, να ολοκληρώσω λέγοντας ότι νομίζω τα κριτήρια που έχουν προβλεφθεί για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα προγράμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, πρέπει να ιεραρχηθούν καλύτερα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς η ασφάλεια της παροχής και η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά θα πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία που θα καθοδηγήσουν την κρατική χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω το διάβημα του εισηγητή και τα σχόλιά του επί του θέματος, διότι σε δύο λεπτά βέβαια μπορεί κανείς να εστιαστεί περισσότερο στα αρνητικά και όχι στα θετικά και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στηρίζουμε βεβαίως την ε, ιεραρχία την οποία αναφέρει για την ε, ε, κατάταξη, δηλαδή ιδίω στην εξοικονόμηση ενεργείας. Δεύτερον, να υπάρξουν ευφύη δίκτυα και να εστιαστούμε σε αυτά και καλύτερη ενσωμάτωση των ανανεωσίμων δικτύων, ιδίω στη Βόρεια Θάλασσα, όπου δεν τονίζεται αρκετά για τα δεκαετή προγράμματα. Επίσης μιλάμε για τις διαρροές διοξιδίου του άνθρακα και όταν θα υπάρξει διασύνδεση μεταξύ της Ευρώπης και των τρίτων χωρών μπορεί να υπάρξει μία τέτοια διαρροή που θα πρέπει να μελετηθεί από την Επιτροπή για να διατυπωθούν οι δέουσες προτάσεις. Και τέλος το βασικό είναι η εντόπιση των κριτηρίων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και το αν άνοιγμα, άνοιγμα της διαδικασίας αυτών των προτεραιοτήτων σε όλους. Διότι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε για αέρια από σχιστόλιθο εφόσον δεν υπάρχει ένα βιώσιμο σύστημα εκμετάλλευσής του. Νομίζω ότι αυτό είναι ανεδαφικό. Και όσον αφορά την ε, ε, ε, αίτηση να το εξετάσει η Επιτροπή, επίσης δεν το θεωρώ σημαντικό. Συμφωνούμε επίσης για το θέμα της προωθήσεως των δικτύων ΣΣΕΣ αλλά ό,τι και να γίνει αυτό δεν πρέπει να είναι η βάρον της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδίως οι λόγοι για την επέκταση αυτών είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν γνωρίζω αν μπορούμε να, να ξέρουμε τι θα γίνει μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιμάς και έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα, ε, σαν ε, ανταπόκριση του Κοινοβουλίου ή ε, την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε να εξετάσουμε τη διαφοροποίηση διότι το εμπόριο ενεργείας δεν είναι δυσμενές εάν λοιπόν θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό το θέμα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προβούμε σε δαπάνες όταν υπάρχει ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον για αυτές τις δαπάνες και μία πρόσθετη αξία για την Ευρώπη. Και ένα από τα θέματα αυτά είναι η διαφοροποίηση, διότι θέλω να τονίσω ότι η αυξημένη διαφοροποίηση και στις πηγές πρέπει να τονιστεί. Δεν θα βρούμε τη χρυσή τομή που θα μας επιτρέψει να κοιτάξουμε ε, αντικειμενικά ποια θέματα πρέπει να τύχουν χρηματοδότηση, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε κάθε τρόπο να προσεγγίσουμε το στόχο αυτό. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Γκιούρκ είναι ο επόμενος που έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. θα ήθελα και εγώ να σας πω ότι θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ ισοσκελισμένη έκθεσή του όπου τίθενται διάφορα θέματα για πρώτη φορά και θέλω να είμαι αισιόδοξο. Θέλω να τονίσω ότι αυτό το μήνα έχουμε διατυπώσει την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ε, στρατηγική για την ενέργεια και τη διαπραγματευόμαστε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμη μία ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτό, αλλά μπορεί να τα αποκτήσουμε στο μέλλον. Ε, ε, επίσης, τροπολογίες μου που αναφέρονται στο θέμα αυτό και θα ήθελα να το θίξω τώρα. Δηλαδή ε, υπάρχουν διάφορα θέματα και ένα βασικό από αυτά είναι η παραδόσεις αερίου από την Ρωσία με το οποίο είχαμε ε, δυσμενείς εμπειρίες στο παρελθόν και χρειάζεται η ε, δημιουργία ενός άξονος από βορρά προς νότο και να βρούμε έναν προσανατολισμό ο, άπαξ και θα έχουμε εφαρμόσει τα προγράμματά μας ε, κατά τρόπον όπως είπε ο κύριος Σιμάνσκι να προχωρήσουμε στους τομείς όπου όντως πρέπει να κάνουμε προσπάθειες. Επίσης οι διαδικασίες αποδοχής. Σχεδόν όλοι μίλησαν για τη διαδικασία αποδοχής και αδειοδότησης. Ε, ε, ε, δεν είναι δυνατόν να χρειάζονται 10 χρόνια για ένα πρόγραμμα για να λάβει μία μία άδεια και επίσης ε, ε, δεν θα μπορέσουν ε, έτσι να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από κοινοτικέ πηγές θα πρέπει και εμείς να συμμετάσχουμε αλλά χρειαζόμαστε για να γίνει αυτό ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς ο κύριος Γκίρεκ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να σταθώ σε ορισμένες έννοιες όπως οι κλιματικές αλλαγές, η ενεργειακή ασφάλεια, πράγματα που αναπτύσσονται στην έκθεση και είναι σημαντικά, διότι δεν μπορεί μόνο η δύναμη της αγοράς να μας οδηγήσει στο να διαμορφώσουμε ένα σύστημα κοινών υποδομών. Πραγματικά δεν θα γίνει έτσι. Δεν μπορούμε μόνο να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς. Χρειάζεται μια σφαιρική θεώρηση, γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε. Επίσης πρέπει να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, πιο συγκεκριμένες. Για το σημείο 5, λόγου χάρη, όπου μιλάμε για το στατικικό ορισμό. Ο εισηγητής μιλά για την ανάπτυξη κάποιων ε, στοιχείων στις τρίτες χώρες. Όμως δεν θα συμφωνήσω με την θεώρησή του. Εδώ μπορεί πραγματικά να αντιμετωπιστεί κίνδυνος διαφυγής αερίων ε, του θερμοκηπίου και διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ το πώς θα παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο όλο ζήτημα μπορεί να αντιφάσκει και με τις διατάξεις της σχετικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κατά νου τις διαφορές μεταξύ ε, των γεωγραφικών ζωνών αναοράριο... ανα και βεβαίω και ανάλογα με τι κλιματικέ αλλαγέ. Άλλε είναι οι συνθήκε στο Νότο και άλλε στην ε, Βόρεια Θάλασσα ή την Βαλτική. Αυτά νομίζω τα ακούσαμε και χθε. Ε, να τα λάβουμε λοιπόν υπόψη. Ευχαριστούμε κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Σόζα Βάγκνερ για την πολύ πλήρη έκθεσή του. Εδώ θέλω να κάνω και εγώ δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα η σημασία της χρήσης των υποδομών ε, φυσικού αερίου της Ιβηρικής Χερσονήσου ε, ως παράγοντα μεταφοράς ε, αυτού του στοιχείου και για την αποθήκευση και για την μεταφορά. Η Ισπανία και η Πορτογαλία διαθέτουν εργοστάσια για την επεξεργασία του αερίου και μπορούν να διευκολύνουν τη διασύνδεση του συστήματος φυσικού αερίου του ευρωπαϊκού επιτρέποντας τη διασύνδεση από τα δικά μας εργοστάσια ως σημείο και για την υπόγεια αποθήκευση και για την ασφάλεια της ε, προμήθειας και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς είναι πολύ σημαντική αυτή η αξιοποίηση. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να συμπεριληφθεί μέσω μιας τροπολογίας είναι ότι γίνεται λόγος για ενεργειακές νησίδες. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να μην ξεχνάμε τα φυσικά, τα από γεωγραφικής άποψης, πραγματικά νησιά. Τα αυτά αυτά νησιά. Εκεί έχουμε τις εξόχως απομακρυσμένες ε, περιοχές, τις ε, ε, Αζόρες, τις Καναρίες νήσους, τη Μαδέρα. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε και από την πλευρά της ενέργειας και της ενεργειακής τους επάρκειας. Αυτά θα ήθελα λοιπόν απλώς να ληφθούν υπόψη. Κατά τα άλλα συμφωνώ πολύ με την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Φανίστελ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να ενώσω τη φωνή μου με τους υπόλοιπους που ευχαρίστησαν τον εισηγητή για την έκθεσή του. Εδώ λοιπόν όντως πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ της διαχείρισης και της παραγωγής αποθήκευσης ή μεταφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι εδώ πρέπει να ε, διδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο η δημόσια κρατική ευθύνη. Έχουμε αρκετά καλά παραδείγματα σχετικά. Η δημοσια κρατικη ευθυνη εχουμε αρκετα καλα παραδειγματα σχετικα γερμανια κατοχώρες, λόγω της ε, τρέχουσας κρίσης έχουν ε, σκεφτεί πώς ε, θα λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτή τη διάσταση. Ως προς τα, την περιφερειακή διάσταση. Μιλήσαμε για το Βορρά, την Ανατολή της Ευρώπης. Ποιος όμως θα επενδύσει στις ανεμογεννήτριες και την αιωλική ενέργεια. Κάποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί. Όμως νομίζω ότι η αγορά μπορεί να ρυθμίσει σε ένα μεγάλο βαθμό τις ανάγκες μας σχετικά με όλα αυτά τα θέματα. Έπειτα για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το σχεδιασμό προγραμμάτων. Νομίζω τα κριτήριά μας θα πρέπει να είναι λίγο πιο σαφή, πιο συγκεκριμένα. Βρισκόμαστε πάντοτε στα όρια μεταξύ των ε, όσων μας έχουν απομείνει από το παρελθόν ε, ως κατάλοιπο και του μελλοντικού στόχου του 10%. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη, ιδίω με διασυνοριακές ανάγκες, να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες επιλογές και για τους σκοπούς της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς μιλάμε για μακροπεριφερειακές περιοχές ή μιλάμε για ευρύτερες περιοχές όπως η Βόρεια Θάλασσα, η Βαλτική. Νομίζω ότι η προσέγγιση αυτή είναι καλή μεν, αλλά θα πρέπει τα αποτελέσματα που θα μπορέσουμε να αντλήσουμε να είναι και αξιοποιήσιμα. Ευχαριστούμε κυρία Τσίκαου. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές μας για την πολύ πλήρη έκθεσή τους. Θα ήθελα να τονίσω την ε, σημασία των εφιών δικτύων και την ε, ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τα ενεργειακά δίκτυα των πόλεων και αναφέρομαι στην κεντρική θέρμανση στην Ευρώπη, ιδίω στα νέα κράτη-μέλη όπου το σύστημα είναι παλιό και χρειάζεται χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσουμε περισσότερο την ενεργειακή αλληλεγγύη και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει ενέργεια σε σωστές τιμές για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κατάλαβα απολύτως αυτό το οποίο ήθελε να πει ο εισηγητής στο 5 ίσως μπορεί να το σχολιάσει πιο εκτενώς και επίσης νομίζω ότι είναι βασικό να τονίσουμε τη σημασία της Μαύρης Θάλασσας και του νοτίου διαδρόμου όσον αφορά τα εφή δίκτυα θα ήθελα να υπάρξει καλύτερη εσωμάτωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εις τα ΕΦΗ δίκτυα μεταφοράς και ενεργείας και να υπάρχει μία αποκέντρωση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Μιλώντας για τις ευφυείς πόλεις και για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα πιστεύω ότι επίσης πρέπει να τονιστεί αυτό το θέμα και θα έπρεπε να βάλουμε στόχο το 2013 και όχι το 2014 για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ο κύριος Βίλα Κουάντρας έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, συνάδελφο Σόζα Βάγνερ ε, για την εξαιρετική του δουλειά. Έκανε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους εγχειρήματα. Έχει καταφέρει να υπάρχει ιδιαίτερη ισορροπία. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι παρά την εξαιρετική του δουλειά, θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες ε, που αποκινούμε την, ε, με ε, τον συντονιστή της ομάδας μου τρεις κατηγορίες ε, τροπολογιών. Πρώτον, για την ενεργειακή αποδοτικότητα θα ήθελα να ε, δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία και για τις επιχειρήσεις και για την ανταγωνιστικότητα. Δεν αφορά μόνο την προσπάθεια ε, μείωσης των επενδυτικών αναγκών η, η, ενέργεια αποτελεί πραγματικά έναν κινητήριο μοχλό για την ανταγωνιστικότητά μας και δεδομένου ότι υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μεγάλο βαθμό στο ενεργειακό μας μείγμα, Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερη ομάδα τροπολογιών, κριτήρια για το ευρωπαϊκό συμφέρον. Έχουμε συμπεριλάβει κάποιες αλλαγές στη δομή των άρθρων και το περιεχόμενό τους. Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ετερογενής, είναι διαφορετικές οι ανάγκες, διαφορετικές οι ιδιαιτερότητες και διαφορετικές οι συνθήκες ε, για την ενεργειακή πολιτική και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και όπου είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για αυτό το πολύ σημαντικό, σημαντικό, το πολύ σημαντικό θέμα των κριτηρίων. Τρίτη ομάδα ε, τροπολογιών αφορά τις άδειες και τις διαδικασίες αδειοδότησης. Εγώ είμαι κάπως ε, επιφυλακτικός σε σχέση με την ε, δυνατότητα ορισμού μια συγκεκριμένης προθεσμίας για τις διαδικασίες αυτές και δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί πραγματικά να ασκήσει επιρροή όσον αφορά την αλλαγή των διοικητικών διαδικασιών στα κράτη-μέλη. Θα ήταν ίσως πιο ρεαλιστικό να ε, επιτρέψουμε την πάροδο 5 ετών ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει την ιδέα μιας διαδικασίας επί επί την βάση του άρθρου 194 της συνθήκης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάπως πιο ρεαλιστικό και επίσης συνάδει περισσότερο με το πρωτογενές δίκαιο. Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι τον εισηγητή και να πω και πάλι ότι είμαι διαθέσιμος να, να ε, βοηθήσω όπως μπορώ. Eh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή, όπως έκαναν και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το σχέδιο έκθεσής τους και νομίζω ότι η έκθεσής του και πιστεύω ότι βάσει του κειμένου αυτού μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάποιες τροπολογίες για να το τελειοποιήσουμε. Ανέφερε ε, ο κύριος Κάριντς, για παράδειγμα, την ιδέα της αποσαφήνισης ορισμένων σημείων στην έκθεση προκειμένου να είναι πιο σαφής. Όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για ε, την ε, ενεργειακή υποδομή, πρέπει να μιλήσουμε για δύο διαφορετικά είδη ενεργειακών υποδομών. Υπάρχει το δίκτυο διανομής όπως υπάρχει και υπάρχουν και μεταφορές. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δύο στοιχεία γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες εχμής σε συνδυασμό με τον τομέα των μεταφορών. Γιατί αν για παράδειγμα ε, το σύστημα ε, των δικτύων δουλεύει αλλά δεν υπάρχει η απαραίτητη τεχνολογία για την υποστήριξη του συστήματος αυτού, αυτό που ουσιαστικά γίνεται ε, είναι ότι δεν, δεν, δεν έχουμε το στόχο της ενεργειακής αποδοτικότητας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η ενεργειακή υποδομή, γιατί και στα δίκτυα ε, διανομής πρέπει οπωσδήποτε, στα, στα δίκτυα παροχής ενέργειας πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται. Ε, τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, πρέπει να είναι και αυτά πιο αποδοτικά στη χρήση ενέργειας. Έχουμε λοιπόν τεχνολογίες εχμής προς την κατεύθυνση αυτή και αυτό σημαίνει ότι πρέπει με τις τεχνολογίες αυτές, τις τεχνολογίες αυτές να τις λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί από αυτές θα προκύψει η τεχνολογική ε, ανάπτυξη, η απαραίτητη για την υποστήριξη των δικτύων αυτών. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βοηθήσει στην ανάπτυξη των ευφυών δικτύων. Ο εισηγητής το γνωρίζει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονιστεί περισσότερο και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνει ήδη. Είναι σημαντικό να τονιστεί ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα, οπότε εγώ θα υποβάλω σχετικώ τροπολογίε, ε, ανάπτυξη δηλαδή μεγάλη κλίμακα προγραμμάτων, για να μπορέσουμε να δούμε το όφελο, τη σχέση κόστου-οφέλου των δικτύων αυτών. Όσον αφορά τώρα την νομοθεσία για τα εφή δίκτυα που σημαίνει προσέλκυση επενδύσεων ε, στον τομέα αυτό, αυτό πρέπει να γίνει πριν από το τέλος του 2011 και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά ε, σημαντικό να αναπτύξουμε υποδομές ε, και για τις μεταφορές. Συγχαρητήρια λοιπόν στον συνάδελφο Σώσα Βάγνερ. Ευχαριστώ. Ήταν μια εξαιρετική έκθεση αυτή την οποία μας παρουσίασε ο συνάδελφος Βάγνερ και είμαστε σε μία περίοδο κρίσεως και τα πράγματα εξελίσσονται ρακδαία. Ε, μετά την Ιαπωνία πολλοί θα αναθεωρήσουν τις πολιτικές ε, των κρατών τους και όσον αφορά την ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν να διατυπώνουμε στην έκθεσή μας και ένα όραμα για το μέλλον ε, βλέπω ότι εδώ δεν τοποθετείται η έκθεση αυτή. Θα πρέπει να αποκομίσουμε και τα συμπεράσματα της κρίσεως του 2008 σχετικά με την παράδοση αερίου, φυσικού αερίου και ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε την έκθεση Βιντάλ Κουάντρας η οποία αναφέρεται σε αυτές μας τις εμπειρίες κατά τρόπον ώστε να απευθύνουμε κάνουμε μία έκκληση στα κράτη-μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν ακόμη στην εφαρμογή ε, των αποφάσεων αυτής της έκθεσης να το πράξουν. Οι χώρες ε, της ε, κεντρικής Ευρώπης είναι πάρα πολύ εκτεθειμένες στις παραδόσεις φυσικού αερίου από τη Ρωσία και μπορεί να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια καλύτερη διασύνδεση μεταξύ Βορρά και Νότου και μεταξύ Σλοβακίας και Ουγγαρίας. Επίσης έχουμε αποφασίσει να, καταστήσουμε, να καταρτήσουμε μια τέτοια σύνδεση. Όσον αφορά τη συνεργασία των κρατών μελών πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και σας ευχαριστώ. Η κυρία Χολ. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω την ε, ε, εφαρμογή αυτής της εκθέσεως και πιστεύω ότι ε, οι τροπολογίες δεν αλλάζουν το πνεύμα της έκθεσης, απλώς ε, περισσότερο εμπλουτίζουν ε, ορισμένες ε, απόψεις. Πιστεύω δε ότι πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την ζήτηση αλλά και την προσφορά και όσον αφορά τα FEE e δίκτυα πιστεύουμε ότι πρέπει να τονίσουμε ότι ο καταναλωτής και ο τελικός χρήστης πρέπει να υποφεληθούν από αυτά τα FEE e δίκτυα και να μην ε, είναι ε, δύσχριστα ε, τα νέα αυτά προγράμματα. Θα πρέπει δηλαδή να προτρέξουμε λιγάκι της, του κανονισμού κατά τρόπον ώστε να εφαρμόσουμε το ταχύτερο δυνατόν το θέμα αλλά συμφωνώ απολύτως με την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριο Σοντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και να του πω ότι είναι βασικό να εξετάσουμε πολιτικά τις υποδομές και καταρχήν θα ήθελα να ορίσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για ενεργειακές υποδομές γιατί νομίζω ότι μιλάμε περισσότερο για διευρωπαϊκά δίκτυα από ότι για υποδομές. Ένας πυρνικός σταθμός είναι μια υποδομή και εγώ θα ήθελα να αναφερθούμε περισσότερο εις ε, τις ε, ενεργειακές εγκαταστάσεις και να ρωτήσω τον εισηγητή τι ε, πιστεύει για το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ποιος είναι ιδιοκτήτης των δικτύων. Μπορεί μια μεγάλη εταιρεία η οποία κάνει επενδύσεις να είναι ιδιοκτήτης των δικτύων διότι δεν νομίζω ότι ο ανταγωνισμός ανταγωνισμός ε, εντός του δικτύου ε, είναι εφικτός εφόσον όλα είναι ρυθμισμένα και δεν υπάρχει ε, ανταγωνισμός. Επίσης επανέρχομαι ποιος πρέπει να θεωρηθεί ιδιοκτήτης των δικτύων και μήπως ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα δίκτυα θα ανήκουν στο δημόσιο και δεν θα μπορούν να εξαγοραστούν από την Κασπρόμι ή κάποιον άλλον. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μία αξιολόγηση και να ξεφύγουμε από την ασάφεια η οποία χαρακτήρισε τις χθεσινές παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν ξέρω ποιος, έχω ένα χαρτάκι εδώ, οπότε παρακαλώ όποιος είναι υπεύθυνος να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή σας, τον κύριο Σόζα Βάγνερ, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι προκειμένου να εξηγήσουμε όλα τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την ενέργεια και τις υποδομές της, ιδίως με, τη, με τα διευρωπαϊκά δίκτυα για την ενέργεια, Είχαμε πολλά θετικά στοιχεία, μια πολύτιμη συνεισφορά από την ακρόαση που οργανώθηκε εδώ χθες. Αλλά και από το σχέδιο έκθεση του συγγετή σα. Ήθελα λοιπόν και εγώ να κάνω κάποιε παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, για τον ορισμό των προγραμμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο. Εδώ θέλουμε να αποφύγουμε τα προκαθορισμένα προγράμματα αλλά περισσότερο να στραφούμε προς αυτά τα οποία κατά την εξέλιξή τους θα προσαρμόζονται στις ανάγκες και με μετρήσιμα κριτήρια τα οποία θα μπορούμε να εντοπίσουμε και να επανακαθορίσουμε. Αυτή τη στιγμή ήδη με τους ιδιοκτήτες των δικτύων ε, που είναι διαχειριστές ε, της ενέργειας συζητούμε καθώς και με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Το λέω αυτό για τον κύριο Οντί. Και αναζητούμε τα κατάλληλα οικονομικά κριτήρια και για την ηλεκτρική ενέργεια και για το φυσικό αέριο. Αυτό βεβαίως θα συζητηθεί με όλους τους ενδιαφερομένους στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί εδώ θα πρέπει να ληφθούν Προφανώ υπόψη. Η ένταξη στην αγορά. Ε, πραγματικά, ε, κύριε Κάρινς, είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και ένας τρόπος είναι ακριβώς να βελτιώσουμε τις υποδομές, η ασφάλεια της προμήθειας. Ένα κριτήριο το οποίο δεν αναφέρεται στην έκθεση του κ. Σόζα Βάγνερ και το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη δική μας άποψη. Σε αυτό έδωσαν έμφαση αρκετοί από τους βουλευτές που έλαβαν το λόγο. Η ασφάλεια της προμήθειας λοιπόν είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για το πώς θα οικοδομήσουμε τις νέες υποδομές. Κυρίως για να εξαλειφθούν οι ενεργειακές νησίδες μεταξύ των χωρών της Βαλτικής ή τη μεταξύ Βόρειας και Νότιας, Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Εκεί υπάρχουν προγράμματα μείζωνος σημασίας για την περιφερειακή συνεργασία, προκειμένου να προχωρήσει η σχετική ενεργειακή προσπάθεια για όσου ακόμη έχουν ενεργειακέ νησίδε, σα διαβεβαιώνω. Έχουμε πάρει την περιοχή τη Βαλτική πολύ σοβαρά και έχουμε θέσει τον δάκτυλο επί τον τύπο όλων των τύπων και προβλημάτων που απασχολούν την περιοχή αυτή. Υπάρχει εδώ ένα μνημόνιο κατανόηση που τουλάχιστον απαριθμεί όλα τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν και έχουμε και ένα εργαστήριο το οποίο μελετά τα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Επίση, μόλι ξεκινήσαμε τι διασυνδέσει με Βορρά και Νότο, δηλαδή να διασυνδέσουμε την Πολωνία με την Τσεχία, την Σλοβακία, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία και να καταφέρουμε να διασυνδέσουμε τελικά τη Βαλτική με την Αδριατική. Τα πράγματα προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα όπως ε, σωστά παρατήρησαν και οι περισσότεροι βουλευτές. Είναι καλές οι ειδήσει. Υπάρχει πολύ καλή διάθεση από πλευράς όλων των παραγόντων οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν προκειμένου να εντοπιστούν αυτά τα προγράμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Προκειμένου να ε, ενοποιηθεί ακριβώ η αγορά και να διασφαλίσουμε την ε, επάρκεια τη ενέργεια και τη προμήθεια. Αυτά είναι τα καλά νέα. Βέβαια υπάρχουν και τα προβλήματα. Χθε τα ακούσαμε. Είναι πολύ σαφέ. Χθε το ακούσαμε. Η αδειοδότηση είναι πολύ ε, χρόνο. Δεν μπορεί να χρειάζεται μια δεκαετία. Είναι απαράδεκτο αυτό και εκεί χρειάζεται στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου. Θέλουμε να υπάρχουν χρονικά περιθώρια και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Βιντάλη Κουάντρα για τα όσα προτείνει. Επίσης η ενιαία θηρίδα ως πρόταση νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση και θα πρέπει να θυμηθούμε και το γερμανικό παράδειγμα του κυρίου Φανίστερο για το πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις ε, διοικητικέ δυσκολίε. Για την χρηματοδότηση θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και οι αρμόδιε εθνικέ αρχέ για να μπορέσουμε να πετύχουμε του στόχου μα. Το συζητούμε μαζί του για να αποσαφηνίσουμε το επενδυτικό κλίμα που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Βεβαίω χρειάζονται ακόμη ευρωπαϊκά κονδύλια για να βοηθήσουμε την όλη προσπάθεια και να εξεύρουμε και καινοτόμα μέσα χρηματοδότηση για τα έξυπνα δίκτυα. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει την ανακοίνωσή τη που σύντομα θα υποβληθεί και εσεί θα λάβετε σύντομα το έγγραφο για να μπορέσετε να τα συζητήσετε και να, τα δει, να δείτε όσα συζητήσαμε σήμερα από το φω ε, αυτή τη ανακοίνωση. Βεβαίω υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για τα έξυπνα δίκτυα, για την αποτελεσματικότητά του και την καλύτερη διαχείρισή του, παρόλο που έχουν γίνει ήδη σοβαρέ προσπάθειε. Σα ευχαριστώ και πάλι για τη δουλειά σα και όλε τι συνεισφορέ. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε και θα φροντίσουμε να έχουμε την κατάλληλη πρόταση μέχρι το τέλο τη χρονιά. Ευχαριστώ. Κύριε Σούζα Μάγνερ, θέλετε να παρέμβετε και πάλι. Ναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για όλα τα καλά σας σχόλια σε σχέση με την έκθεσή μου. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου ετέθησαν από την κυρία Τικάου σε σχέση με το θέμα της διαρροής του άνθρακα στην ε, παράγραφο 15 της έκθεσης. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο δεν αναφέρεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει να κάνει με τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Αυτό που ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να εξετάσει τα προβλήματα που προκύπτουν από το ζήτημα αυτό και να προσπαθήσει να ε, υπάρξει ένας ε, μηχανισμός για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τη διαρροή αυτή ή να ε, δούμε πώς εφαρμόζεται η οδηγία σχετικά με το θέμα αυτό. Σε σχέση με τα σχόλια του κυρίου Οντή, πολύ ορθώς έθεσε το ζήτημα της ιδιοκτησίας των δικτύων και όλων των σχετικών στοιχείων. Άλλωστε αυτό αναφέρθηκε και στη χθεσινή συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες. Βέβαια, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές απαντήσεις σε αυτό το θέμα. Το κάθε κράτος μέλος ε, αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό με το δικό του τρόπο. Πολλές φορές έχουν προσπαθήσει κάπως να διαφοροποιήσουν τους μηχανισμούς μεταφορών, άλλες φορές δεν έχουν καταφέρει να βρουν την καλύτερη λύση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιες λύσεις. Το θέμα των ενεργειακών νησίδων, το θέμα της αποδυτικότητα των ε, αγορών, της ενιαίας αγοράς, όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα όταν φτάσουμε στη συζήτηση για τις τροπολογίες να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Η προθεσμία είναι σε μερικές μέρες και θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε σε αυτό και να το εξετάσουμε υπό το φως όλων των ε, συνεισφορών που θα στείλουν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους πάρα πολύ και ελπίζω να εξακολουθήσουμε να να εξακολουθήσω να στην υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες ε, είναι σύντομη διότι θα πρέπει να έχουμε ψηφίσει μέχρι τις 26 Μαΐου. Οπότε ε, θα περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την ανάλυση των επιλογών για την ε, κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση των κινδύνων διαρροής ε, άνθρακα. Ε, άρα ο κύριος Καρβάλιο θα κάνει την παρουσίαση, η κυρία Καρβάλιο θα κάνει την παρουσίαση αντί για τον εισηγητή που δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η κυρία Τζορντάν μου ζήτησε να παρουσιάσει την ε, έκθεσή της και θα κάνω μία σύντομη περίληψη. Υπάρχουν πέντε θέματα. Το πρώτο είναι ότι η συγγήτρια θέλει να περιγράψει πού βρισκόμαστε με το στόχο μας του 80% αν είμαστε ή όχι στο σωστό δρόμο δεδομένης της οικονομικής κρίσης και να τονίσει το μακροπρόθεσμο στόχο του 2050. Επίσης ε, ε, θέλει να, μη, να ε, αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των ενεργειακών δικτύων και του προγράμματος πλαισίου και να ε, αξιολογήσουμε τα υπέρ και τα κατά του να προχωρήσουμε πέραν του 20% μειώσεως για να δούμε ε, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μία μονομερή κίνηση για μείωση πέραν του 20% και ποια θα είναι τα υπέρ και τα κατά για την Ευρώπη. όσον αφορά το θέμα, τέταρτο θέμα για την διαρροή ε, διοξιδίου του άνθρακος υπάρχει για την βιομηχανία και ο συγγήτρια πιστεύει ότι η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρά είναι αισιόδοξη και τέλος όσον αφορά τις περαιτέρω δυνατότητες και τις προκλήσεις η συγγήτρια θεωρεί ότι δεν πρέπει να μιλάμε για στόχους αλλά να τονίσουμε τους μηχανισμούς και τα εργαλεία για να τους επιτύχουμε για, κατά τρόπον ώστε τουλάχιστον να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς δηλαδή να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τέλος η συγγήτρια σας καλεί όλους στην ακρόαση που θα γίνει αύριο 9 με 12.30 εις ε, την αίθουσα John 4Q1 ε, με μία παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά που απασχολούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ που μας βοηθήσατε σήμερα και ο κύριος Τζαντούλας είναι ο πρώτος ο οποίος θα λάβει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως έχουμε αυτή τη συζήτηση με τον εισηγητή ε, με επικοδομητικό ο κύριος Ζαντό, με συγχωρείτε, έχει το λόγο και βλέπουμε ότι μπορούμε ε, να ε, είμαστε πιο ευέλικτοι για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις διότι οι φιλόδοξοι στόχοι μας θα μπορούσαν να τα στρέψουν όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία και από την άλλη πλευρά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν πρέπει να, να παραβλέψουμε τις ε, διαρροές διοξιδίου του άνθρακος. Πιστεύω λοιπόν ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να είναι ε, πολύ ρεαλιστική, πράγμα το οποίο μας οδηγεί στο να συζητήσουμε και να προτείνουμε ορισμένες τροπολογίες σχετικά με την έκθεση. Τύπικα όταν στην έκθεση μας λέγεται ότι η οδός το cost effective pathway είναι να παραμείνουμε στο 20% δείχνει ότι δεν ε, συνάδει με τις εργασίες που έχει αναλάβει αφενός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σχετικά με τις ανακοινώσεις που έχει ήδη καταρτήσει και τους εμπειρογνώμονες άρα θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Δεύτερον, λέγεται στην έκθεση ότι σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες η πολιτική η τωρινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε ήδη να οδηγήσει σε ε, μετακινήσεις και μεταθέσεις ε, των ε, εργοστασίων σημαντικών. Καμιά όμως σοβαρή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν επιβεβαιώνει αυτό το κίνδυνο. Άρα όσον αφορά τη διαρροή του διοξιδίου του άνθρακος πρέπει να δούμε τι αναγράφεται. Είπαμε ε, και εμείς ότι όταν υπάρχει κίνδυνος διαρροής θα πρέπει να προστατευτεί ο τομέας αυτός κατά τρόπον ώστε να παραμείνει στην Ευρώπη και να προσαρμοστεί στην ενεργειακή πραγματικότητα. Τέλος λέγεται ότι ορισμένες ε, ε, επιχειρήσεις ε, θα πληρώσουν πολύ ακριβά όλες αυτές τις προσαρμογές. Θυμάστε ότι για επιχειρήσεις σαν την Ασελόρο Μιτάλ υπήρχε ε, ε, ένα κέρδος 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Λαφάζ εκατομμύρια ευρώ και βλέπετε ότι οι επιχειρήσεις έχουν κερδίσει μέχρι στιγμής ε, μέχρι και υπερβολικά από την ευρωπαϊκή πολιτική. Οπότε θέλουμε να συμβάλλουμε κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ένα γραφείο το οποίο ε, βοηθά τις ε, ε, επιχειρήσεις που κινδυνεύουν αλλά μην παραβλέπουμε ότι παράγουν οι εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο που αποδεικνύουν ότι η κλιματική φιλοδοξία είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Η κυρία Ματίας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με, το, με όσα είπε ο συνάδελφος μόλις τώρα. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουμε σε κάποιους καλούς συμβιβασμούς και γι' αυτό πρέπει να εγκρίνουμε ε, μία επικοδομητική προσέγγιση. Γιατί εννοώ επικοδομητική να μην λέμε μόνο τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά να δούμε και τι μπορούμε και εμείς να προτείνουμε ως Κοινοβούλιο από τη δική μας πλευρά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Αν θέλουμε πράγματι να ασκήσουμε επιρροή ε, στην ε, νομοθεσία που εξετάζει τα ζητήματα αυτά της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να έχουμε αυτή την επικοδομητική προσέγγιση για να μπορέσουμε ακριβώς να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. Το έγγραφο λοιπόν για την κίνηση προς μια πιο ανταγωνιστική οικονομία μέχρι το 2015 είναι ένα από τα έγγραφα που θα πρέπει να τα σκεφτούμε εδώ. Ε, ιδίω σε σχέση με τις ευθύνε που έχουμε αναλάβει για τον περιορισμό των εγχώριων εκπομπών, των ευρωπαϊκών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε μια ισορροπία και μεταξύ αυτών των υποχρεώσεων και των περιορισμών που μας επιβάλλονται και των στόχων που έχουν τεθεί. Επίσης θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας ως ε, συνήθως. Business as usual δεν μπορεί να είναι η αρχή που θα μας ε, διέπει πλέον. Πρέπει εδώ να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να λάβουμε κάποια μέτρα και να προστατεύσουμε αυτό το βιομηχανικό κλάδο έχοντας υπόψη και τις απαραίτητες προσαρμογές που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ προκλήσεις τη βιωσιμότητα και των κλιματικών αλλαγών και άλλων που ήδη αναφέρθηκαν. Στην πραγματικότητα, δεν είναι ότι ζητάμε πολλά ή περισσότερα. Τα είχαμε συζητήσει από το 2008 επί Γαλλικής Προεδρίας. Είχαμε αναλάβει και είχαμε προχωρήσει σε μια σειρά από συμφωνίες και πρόβλεψη μέτρων που δεν ήταν αρνητικές, ίσα ίσα ε, για, τα για το βιομηχανικό κλάδο ιδίω, ο πρόεδρο Σαρκοζή είχε αναλάβει συγκεκριμένε ευθύνε. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε αυτέ τι υποσχέσει. Για ε, το συνάδελφο λοιπόν να πω ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να φτάσουμε σε επικοδομητικέ συμβαστικέ λύσει και μια προσέγγιση εύστοχη ώστε να διευκολύνουμε και το βιομηχανικό τομέα και να επιτύχουμε όλου του στόχου που όλοι οι συναδελφοί προανέφεραν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μετσάρος. Ευχαριστώ το 2008 αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μία εκστρατεία για την μείωση των εκπομπών και τώρα βλέπουμε ότι θέλουμε να προβούμε σε μία μείωση μέχρι και 30%. Έκτοτε όμως άλλαξε η κατάσταση, υπήρξε μία χρηματοοικονομική κρίση η οποία επηρεάζει και τους ε, προϋπολογισμούς της Ευρώπης και τις δυνατότητες δαπανών. Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ε, να ε, καταπολεμήσει το θέμα των εκπομπών και πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τουλάχιστον τη μείωση των 20% και ενδεχομένως να επιστήσουμε και μία μείωση 30%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να εστιαστούμε στις περιοχές όπου υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε την κατάσταση γιατί ξέρουμε ότι τώρα η μείωση του 20% συνεπάγεται λιγότερα έξοδα από ό,τι νομίζαμε και άρα πρέπει να ξανασκεφτούμε και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Οι προϋποθέσεις δεν υφίστανται ακόμα ακόμη για μία μείωση 30% αλλά πρέπει να επιφυλαχθούμε για το μέλλον και να προετοιμαστούμε για να προβούμε στη μείωση αυτή όταν θα υπάρχουν οι αναγκαίες συνθήκες. Και ε, κατόπιν των γεγονότων της Ιαπωνίας πιστεύω ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα χρειαστεί να αναθεωρήσουν την πολιτική τους διότι βλέπουμε ότι ε, πρέπει ε, να δούμε και εμείς και να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των στόχων γιατί δεν έχουμε ε, επαρκείς δυνατότητες να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και θα χρειαστούμε διεθνείς συνεργάτες. Ο κύριος Γκίρεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συνάδελφοι, έχουμε να εξετάσουμε εδώ μια έκθεση ιδιαίτερα ισόρροπη για ένα θέμα πολύ ευαίσθητο για τον περιορισμό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ δεχόμαστε πιέσεις από την πλευρά των ε, ομάδων ασκήσεως πίεσης και όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή μπορούν να καταλάβουν τις επιπτώσεις ενός πακέτου μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές που έχει επιβληθεί αυθαίρετα. Σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα την έκθεση τώρα. Να σταθώ στην παράγραφο 4 όπου μιλάμε για μείωση κατανάλωσης ε, κατά 20%. Δεν υπήρξε τέτοια συμφωνία εξ όσων θυμάμαι. Γίνεται λόγος για τον στόχο του 2020 αλλά και για αύξηση της αποδοτικότητας ε, κατά το 20%. Ε, δεν είναι το ίδιο αυτό με την με τον περιορισμό της κατανάλωση κατά 20%. Εδώ λοιπόν είναι λανθασμένος ο ορισμός. Επίσης το να λέμε ότι θέλουμε να πετύχουμε κάποιους στόχους ε, μέχρι το 2020, ναι, είναι κάτι για το οποίο σίγουρα υπάρχει πολιτική βούληση. Όμω, στον παράγραφο 16 θα πρέπει να πούμε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα ότι στην περίπτωση οικοδόμηση νέων εργοστασίων για την επεξεργασία του φυσικού αερίου θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα νέα κριτήρια. Και το ίδιο και για τα εργοστάσια με την ε, που λειτουργούν με βάση τον άνθρακα και την ε, παγίδευση των αερίων του θερμοκηπίου και των διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα, να ευχηθώ καλή τύχη στην εισηγητρία. Εύχομαι να επιστρέψει σύντομα. Και κυρίως να την ευχαριστήσω για τις ε, πλήρεις μεθόδους εργασίας που χρησιμοποίησε. Τέλος πάντων που ξεκίνησε να χρησιμοποιεί πριν να στενήσει. Ελπίζω, ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε την εξέταση του όλου θέματος κατά τον ίδιο τρόπο. Να πω ότι την έκθεση αυτή τη βρίσκω λίγο απεσιόδοξη. Εάν δω πιο πρόσφατες εκθέσεις όπως αυτή που η γερμανική κυβέρνηση ζήτησε από το Ίδρυμα του Πότσταμ πριν από δύο-τρεις εβδομάδες ήταν λίγο πιο αισιόδοξη και μάλιστα κατά διάφορους τρόπους. Από επιστημονικής άποψης λόγου χάρη, οι αναφορές της έκθεσης αυτής είναι αρκετά αξιόπιστες και το Ίδρυμα αυτό έχει πολύ καλή φήμη. Εάν δεχτούμε λοιπόν την ανάλυση τους και την ανάλυση της ανακοίνωσης και του κυρίου Έτιγκερ και του κυρίου Έρεμπορντ, για την ενεργειακή αποδοτικότητα, θα δούμε ότι ο πιο αποτελεσματικό ω προ το κόστο τρόπο να πετύχουμε αυτό το στόχο είναι τη μείωση του 20% στο 2020 να την αντιληφθούμε ως μια ανεπαρκή προσπάθεια. Η βιομηχανία θα πρέπει να επενδύσει περισσότερα με πιο εξυγχρονισμένα μέσα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει μέχρι το 2050 να μην αναζητούμε μία καμπύλη, αλλά μία ευθεία γραμμή και για τις επενδύσεις και για το κόστος, ε, για πολλούς λόγους. Ε, ήδη εκδόθηκαν, ε, δημοσιεύτηκαν δύο έγγραφα για το θέμα αυτό και αυτά μπορεί να φαίνονται περίεργα, όμως η βιομηχανία γνωρίζει καλά ποιο είναι το μέτωπο που θα εξελιχθεί αυτή η μάχη και γνωρίζει και ποιε είναι οι δυνατότητε. Εάν κοιτάξουμε την αγορά σε διάφορου τομεί, λοιπόν, για τα οχήματα λόγω χάρη ή για τα φορτηγά, θα δούμε ότι οι πελάτε, οι καταναλωτέ αγοράζουν οχήματα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια το ίδιο και για τι συσκευέ ε, που χρησιμοποιούνται στα νοικοκυριά των πολιτών. Έχουμε ξεθαύμαστε ε, επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα. Το ίδιο ισχύει και για τα κτίρια. Η αγορά κινείται. Το οικονομικό επιχείρημα για τη σημερινή κατάσταση είναι ότι το να στρεφόμαστε μόνο προς την οικονομική κρίση ε, μας οδηγεί και στο εξή συμπέρασμα. Είναι πολύ πιο φθηνές επενδύσεις τώρα, άρα μπορούμε να ανεβάσουμε τις φιλοδοξίες μας για την επίτευξη των στόχων για την ανταγωνιστικότητα. Το θέμα αυτό το βρίσκω πολύ σημαντικό, ιδίως εάν κοιτάξουμε σφαιρικά την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχει και μια παρατήρηση στην έκθεση Hildegard για τις κεφαλογικές επενδύσεις στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα ή την Ινδία. Βάσει των τελευταίων στατιστικών δεδομένων, η Ευρώπη επένδυσε 19% ενώ η Κίνα 45%. Αυτό σημαίνει ότι το να προσθέσουμε στο 19, μια μισή ποσοστία μονάδα για να περάσουμε από το 19 στο 20 κάτι, είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τις μισές επενδύσεις από το ΑΕΠ, πολύ περισσότερα για να συναγωνιστούμε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Κίνας ή της Ινδίας που έχουν περίπου 40%, η Νότια Κορέα 30% και η Ευρώπη είναι 19%. Είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Είναι πολύ ανησυχητικό το στοιχείο. Δεν είναι λοιπόν μόνο το κόστος ένα πρόβλημα, αλλά και ο χρόνος. Ιδίω για την βιομηχανία και από άποψη οικονομικής. Επίσης, σήμερα πλέον έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση και αυτό το επεσήμανε και Euroelectric με πολύ εύγλωτο τρόπο. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου κινδυνεύουμε με το, από κατακαιρματισμό της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς, ενώ αντιθέτως αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολύ περισσότερη εσωτερική ρύθμιση στην εσωτερική αγορά ενέργειας και πολύ περισσότερες κοινέ προδιαγραφές και κοινή δράση. Μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη συγκυρία. Γνωρίζουμε ότι κατακαιρματισμός ισοδυναμεί με κόστος, με απώλεια θέσεων εργασία. Για τη διεθνή διάσταση έθιξα νομίζω εν μέρει το τι συμβαίνει ε, από την άποψη των επενδύσεων, σημαντικό θα είναι να δούμε και το πενταετές κινέζικο πρόγραμμα, να δούμε τι κάνουν στον τομέα αυτό. Ο τρόπος που επενδύουν ε, στις νέες αγορές, τα νέα τεχνολογικά μέσα, αυτά που ονομάζουμε εμεί πράσινη τεχνολογία, ενώ εκείνοι τα αποκαλούν απλώς νέα τεχνολογία ή αποτελεσματικές προς το κόστος τεχνολογία, αυτό είναι ένα εκπληκτικό στοιχείο αν το σκεφτείτε. Τι κίνδυνο αντιμετωπίζουμε λοιπόν στην Ευρώπη, σκεφτείτε το, εάν δεν αναλάβουμε ηγετικό ρόλο σε αυτήν την περιοχή. Δηλαδή, στην αγορά, στη βιομηχανία, σε αυτούς τους κλάδους, δεν έχουμε ηγετικό ρόλο. Η Κίνα πέρασε στην αιωλική ενέργεια από μηδέν στο 50 περίπου 100 στην αγορά της. Και αυτό ισχύει και για το φυσικό αέριο και για άλλες ενέργειες που δεδομένης της σημερινής κατάστασης και όλων όσων συζητούμε σε αυτή την Επιτροπή και μόλις συζητήσαμε χθε. γίνονται ακόμη πιο σημαντικά υπό το φως και των όσων μας είπε ο Επίτροπος Έτιγκερ. Άρα λοιπόν τον ηγετικό μας ρόλο στις τεχνολογίες αυτές τον διαθέτουμε μεν, αλλά δεν τον αξιοποιούμε. Τον είχαμε κάποτε και τώρα δεν τον έχουμε πια και αυτό μας ανησυχεί βαθιά για το σύστημα ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπής. Εδώ η δυνατότητα μεταφορά των μη χρησιμοποιημένων δικαιωμάτων και μετατροπή του σε κεφάλαια θα μπορούσε να ε, χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις. Δείτε ποια είναι τα κέρδη που μπορούμε να αποκομίσουμε και ας σκεφτούμε ότι δεν είναι να μένουν ε, και να κάθονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις ακριβώς οι ίδιες εταιρείε που έχουν τέτοιους τραπεζικούς λογαριασμούς ανησυχούν για τη διαρροή του άνθρακα. Να τα σκεφτούμε λίγο αυτά. Υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία που μας λένε ότι σε διάφορους τομείς υπάρχουν εταιρείε που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο εργασίας. Να χρησιμοποιήσουν λοιπόν αυτά τα κονδύλια για επενδύσεις. Νομίζω ο κίνδυνος από την διαρροή του άνθρακα είναι πολύ πιο περιορισμένος εάν ε, ενισχύσουμε τα συστήματά μας. Διότι αν οι εταιρείε τα κέρδη τους τα κρατάνε στην Ευρώπη αντί να τα διασκορπίζουν εκτός, Πολλά θα είχαμε να κερδίσουμε. Ιδάλω, νομίζω ότι καταλήγουμε σε μια ηρωνία που... τραγική ηρωνία που θα ήταν καλό να τη σκεφτούμε. Και όσα είπε η κυρία Ματίας είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για μέτρα προσαρμογής βάσει κάποιου δασμού ή φόρων και σε σχέση με τα σύνορα της εσωτερικής αγοράς. Όταν συνεργαστήκαμε και συζητήσαμε την ε, οδηγία για τα χημικά, το REACH, είχαμε ξαναέρθει στα θέματα αυτά. Η Βρετανική κυβέρνηση, θυμόμαστε ότι είχε εκφράσει την ε, συμπάθειά της για όλα αυτά τα θέματα μένα, αλλά ποτέ δεν κατέληξε σε συγκεκριμένα μέτρα. Ε, θέλουμε λοιπόν κάτι αποτελεσματικό και για την αγορά. Και η στιγμή να προχωρήσουμε είναι τώρα. Έχουμε τις απαραίτητες τεχνικές, έχουμε τα μέσα, έχουμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ελπίζω λοιπόν ότι με τους άλλους και όδους εισηγητές θα αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό που έχουμε σε αυτό το, σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Κυρία Τσίκαου. Uh, uh, uh, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να, ευχαριστήσω τους συναδέλφους, την εισηγήτρια, πρώτα απ' όλα, και θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία όσον αφορά την μείωση των εκπομών αερίων θερμοκηπίνου ώστε να μπορέσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια να σημειώσει προόδου σε σχέση με τις δεσμεύσεις της για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Παράλληλα, Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην προσπάθεια αυτή της μείωσης των εκπομπών διοξιδίων του άνθρακα να τονίσουμε ιδιαίτερα την ενεργειακή αποδοτικότητα στον τομέα των μεταφορών αλλά και στον τομέα, για παράδειγμα, ε, της στέγασης των κτηρίων ε, στον οποίο δεν έχουν κάνει πολλές προσπάθειες τα κράτη-μέλη σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια, για παράδειγμα. Δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες προσπάθειες και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επόμενο ε, χρηματοοικονομικό ε, πλαίσιο να ληφθεί υπόψη αυτό το πρόγραμμα δημιουργίας εφιών πόλεων. Γι' αυτό ακριβώς ε, και τα ευφυή δικτύα είναι πάρα πολύ σημαντικά, εξίσου σημαντικά και θα μπορούσαμε να αναμίξουμε την ενέργεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που, ενέργειας που αποτελεί μια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που λαμβάνει χώρα σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο και θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που θα να, θα μπορούσε να μεταφέρει και να διαθέτει ε, σε τοπικό επίπεδο ενέργεια που έχει προέλθει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να υπάρξει και η απαραίτητη υποδομή για τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία θα μπορέσουν και αυτά να συνεισφέρουν στη μείωση των εκπομπών διοξιδίων του άνθρακα που, προ, που, που εκλεί ο τομέας των μεταφορών. Αυτά τα σημεία λοιπόν θα ήθελα να θέσω. Η ενεργειακή αποδοτικότητα ειδικότερα στον τομέα των κτηρίων ε, και έχουμε πολλή δουλειά σε αυτό το τομέα και η ενεργειακή αποδοτικότητα στον τομέα των μεταφορών. Με ιδιαίτερη έμφαση στην ε, ολοκλήρωση των προγραμμάτων των ε, ηλεκτρικών οχημάτων στο πλαίσιο των εφιών ε, δικτύων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι νέες πηγές ενέργειας. Ο κύριος Ρόντε. Συγγνώμη. Καθυστέρησα λιγάκι, λέει ο κύριος Γκρότε αλλά υπάρχει και μία συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος που συζητούνται τα ίδια θέματα, οπότε πρέπει να είμαι πανταχού παρών σήμερα. Το 2008 άρχισε να ισχύει το πακέτο το ενεργειακό και νομίζω ότι η μείωση του, σε, σε 20, κατά 20% μέχρι το 2020 είναι μια καλή ιδέα. Αν συμμετέχουν και όλες και άλλες χώρες από άλλα μέρη του κόσμου θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο 30%. Τώρα πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το 30%. Πρέπει να δούμε τι τακτική θα ακολουθήσουμε για να γίνει αυτό. Γιατί το κλίμα δεν έχει να κάνει μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι χρειάζονται συζητήσει και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης πρέπει και εκείνη να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες διπλωματικής φύσεως παρά το γεγονός ότι η πάτη εκπρόσωπός μας. Ε, ε, καταλαβαίνω ότι έχει και άλλες πολύ σημαντικές υποχρεώσεις. Πρέπει όμως και το θέμα αυτό το ενεργειακό να είναι τμήμα της ατζέντα της και να προσπαθήσει να το προωθήσει σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε αναπτύξει φιλόδοξα κριτήρια. Στην Κανκούν μιλήσαμε για 30%. Θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει και στο 60 ή 70%. Ούτως ή άλλως δεν καταλήξαμε πουθενά. Δεν είναι όμως το συμπέρασμα ε, και η κατάληξη της ε, ε, διάσκεψης που, πρέπει να, που θα μας λέει τι θα κάνουμε. Πρέπει να υπάρξει μια βιομηχανική πολιτική οικολογική. Η, η κυρία Εκ μόλις μίλησε για αυτό το θέμα. <coughs> Νομίζω ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε από τη μία, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε και τη τελική μάχη. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους και να μιλήσουμε για την αύξηση του, του μεριδίου ε, της, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 40%. Υπήρχε ένα σφάλμα ήδη από την αρχή, δεν μπορούμε να μιλάμε για ενεργειακή κατανάλωση. Καλό ε, θα ήταν, μας είπαν, να μιλάμε κυρίως ε, για ενεργειακή αποδοτικότητα, για λιγότερο ενεργοβόρες οικιακές συσκευές για παράδειγμα, συσκευές γενικότερα. Θα έπρεπε λοιπόν να θέτουμε στόχους οι οποίοι να μην, είναι στο, να μην είναι στο περίπου, να είναι πολύ συγκεκριμένοι, να γνωρίζουμε ε, σε ποια προθεσμία συγκεκριμένη θέλουμε να έχουμε επιτύχει ένα αλφα επίπεδο ενεργειακής αποδοτικότητας, η διαρροή του άνθρακα για παράδειγμα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που έχουν ε, αυτό το πρόβλημα και έχουμε λάβει και μέτρα. Στην αρχή είχαμε καταφέρει το έμεσα κόστος στο τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ε, να οδηγεί σε κάποια πλεονεκτήματα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση που θα εγκρίνουμε, αλλά και στην Επιτροπή Περιβάλλοντο νομίζω πρέπει να το θέσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να έχουμε και χρόνο να αποφασίσουμε 20%, 30% και να υπάρχουν και συγκεκριμένα κίνητρα για να φτάσει το θέμα, να προωθήσουμε το θέμα και στην κοινή γνώμη. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ πώς θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, γιατί το κλιματικό, ε, το ενεργειακό πακέτο ας πούμε δεν το ε, γνωστοποιήσαμε πολύ καλά στην κοινή γνώμη. Ε, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πούν την άποψή τους γιατί πέρασε το, πράγμα σε, πέρασε το θέμα σε πρώτη ανάγνωση. Αυτή τη φορά όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να πάρουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τους τομείς στους οποίους μπορούμε να προοδεύσουμε και επιμένω σε αυτό, ειδικότερα στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσουμε προόδους σημαντικές. Η Επίτροπος μίλησε χτες ε, για 40% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020. Νομίζω ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο και νομίζω ότι αυτό συνάδει και με τη στρατηγική για το 2020 γιατί θα μπορέσουμε έτσι να δημιουργήσουμε και νέες θέσεις απασχόλησης. Διότι ο μεγαλύτερος εργοδότης ε, είναι ο τομέας της ενέργειας, ε, τουλάχιστον στη Γερμανία. Έχουμε κάθε μέρα προβλήματα διανομής ορισμένων προϊόντων. Δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια πραγματική βιομηχανική και οικολογική πολιτική. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να εξετήσουμε το CDM και την εφαρμογή του, να δούμε αν δηλαδή τέτοια μέσα μπορούν να επιτύχουν. Είναι κάτι που θα ήθελα επίσης να διερευνηθεί και να αντικατοπτρίζεται στην έκθεση αυτή. Και τέλος, πιστεύω ότι δεν πρέπει απλώς να καθορίσουμε στόχους και μετά να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα, αλλά ε, ό,τι έχει αποφασιστεί για το 2008 να διασυνδεθεί επίσης, δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τη μείωση κατά 20% και να μην ξεχνάμε ότι τελικά πρέπει να φτάσουμε σε πολύ πολύ σημαντικότερη ε, μείωση για να υπάρξει μείωση κατά δύο βαθμούς. Αυτό χρειάζεται. Ε, άρα ποιες πολιτικές αποφάσεις θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν εκεί. Ποιες είναι οι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα ε, εμποδίσουν να επιτύχουμε το στόχο μας. Διότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλη την Ιφίλιο, υπάρχει διεθνής ανταγωνισμός και αυτό το οποίο ε, ίσως ε, υποτιμούμε δεν πρόκειται μόνο για μία μάχη για τη μείωση κατά 20 ή 30% αλλά μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης, για το μέλλον της Ιφιλίου και του πλανήτη μας. Αν θέλουμε δηλαδή να προχωρήσουμε και να επενδύσουμε σε πράσινη τεχνολογία και αν είναι σκόπιμο να δημιουργήσουμε με τέτοια πολιτική την, ε, τις θέσεις εργασίας και την ευημερία αντί να μας φύγουν όλες ε, οι βιομηχανίες και να μείνουν όλοι άνεργοι. Δηλαδή το να μειώσουμε μειώσουμε κατά 2% του 2 βαθμούς τη θερμοκρασία και να μας φύγουν όλοι δεν έχει κανένα νόημα. Άρα θα ήθελα αυτό το θέμα να συζητηθεί και προσκαλώ όλους τους συναδέλφους σε μια τέτοια συζήτηση. Ευχαριστώ. Και τώρα σαν πρόεδρος θα ήθελα να σας πω ότι ε, πρέπει στις διαβουλεύσεις να υπάρξει επαρκής χρόνος διότι και εγώ αντιμετωπίζω το θέμα ακριβώς όπως και εσείς δηλαδή πρέπει να δούμε τι θέλουμε πώς θα προχωρήσουμε να κάνουμε σωστά τις διαβολεύσεις γιατί μετά δεν θα μπορούμε να διορθώσουμε αυτά που έχουν γίνει ο κύριος Φόμποντα. ευχαριστώ θα είμαι σύμφωνος γιατί συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ε, πρέπει να σας πω ότι για να βρούμε και να πετύχουμε πετύχουμε τους στόχους μας χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την, ε, τις βιομηχανίες και τις θέσεις εργασίας, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλές βιομηχανίες προσπάθησαν να μειώσουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τις εκπομπές και ε, θέλουμε να έχουμε και πιο μεγαλεπίβουλους ε, στόχους αλλά έχουμε ασθενή διαπραγματευτική θέση και αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις βιομηχανίες μας. Πρέπει λοιπόν κατά μέσον όρο να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Δεν θα το επιτύχουν όλοι αλλά ε, τουλάχιστον κατά μέσον όρων, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή τη συζήτηση <clears throat> και να μπορέσουμε να διδαχθούμε και από την τραγική κατάσταση της Ισπανίας. Θα πρέπει λοιπόν, της ε, Ιαπωνίας με συγχωρείτε. Όντως θα πρέπει να αυξήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και επίσης τα θέματα που ανέφερε η συνάδελφος Τικάου. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε δεσμευτικούς στόχους αλλά η Επιτροπή θα πρέπει να προτραπεί ε, να ε, διατυπώσει στόχους πριν γίνουν υποχρεωτικοί για τα κράτη-μέλη και να αυξήσουμε ε, την ε, χρήση των ανανεωσίμων πηγών ενεργείας, να μειώσουμε τις ε, εκπομπές αλλά να εξασφαλίσουμε και τις θέσεις εργασίας και τις σωστές μεταφορές. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη διότι τα, ε, αν κοιτάξουμε τα προγράμματα που αποφασίστηκαν την περασμένη εβδομάδα βλέπουμε ότι ζητάμε πολύ λιγότερα από τις μεταφορές από, ότι, από τη βιομηχανία πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό για να διατηρήσουμε τις βιομηχανίες αυτές στην Ευρώπη και γι' αυτό συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Γκρότε. Η κυρία Χέρτσογκ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι στην Επιτροπή μας όλοι συμφωνούν με το στόχο ότι πρέπει να επιτύχουμε το 20% και το πέρα του 20% και επίσης νομίζω ότι όλοι υποστηρίζουμε την αρχική μας ιδέα ότι ο στόχος πρέπει να είναι σφαιρικός και όχι μόνο τοπικός γιατί το διοξίδιο του άνθρακα μέσω του αέρα κυκλοφορεί παντού. Έχουμε πολλή δουλειά. Πρώτα απ' όλα Πρέπει να διατηρήσουμε την απόφασή μας ότι προς τα εκεί θα κινηθούμε και ελπίζω να μπορέσουμε να ε, συνεχίζουμε να δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε πιο αποδοτικούς ενεργειακά ε, μηχανισμούς ε, και ε, κινητήρες. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αναφερθούν ορισμένα πράγματα σε σχέση με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Μέχρι το 2050 η, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί κατά 40%, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τώρα που είμαστε το 2011, ένα επιπλέον άτομο θα χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια κάθε μέρα. Δηλαδή, τα ορυκτά ε, καύσιμα ε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που θα μπορούσε να επιληθεί για παράδειγμα από, ε, την, από, με, τα, ηλεκτρικά οχήματα τα οποία είναι, είναι επίσης πολύ σημαντικό να τα σκεφτόμαστε. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η βασική συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εξή. Κάποιες χώρες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, κάνουν ό,τι μπορούν, ενώ άλλες περιοχές, όπω η δικιά μου για παράδειγμα, που δεν είναι η μόνη, έχουν καθιστορήσει πάρα πολύ. Οπότε οι ασυνέπειες ε, τη επίτευξης των στόχων αυτών είναι τεράστιες. Αν ε, πάει κανείς για προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία και δεν μιλούσε για αυτούς τους στόχους, θα είχαν τις εκλογές. Όμω, αν οι πολιτικοί σε κάποιε περιφέρειες, όπω τη δική μου, α πούμε, μιλούσαν για το στόχο αυτό, ενδεχομένω πάλι να έχαναν την, τις εκλογές. Οπότε αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένας ένα από τα βασικότερα πράγματα, από τα πιο εύκολα πράγματα να επιτύχουμε για να υπάρχει συνέπεια, ε, συνοχή στις προσεγγίσεις ε, έναντι των Ευρωπαίων πολιτών, Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τεράστια ε, ε, ευθύνη και εμείς έχουμε ευθύνη και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς γενικότερα να μην εγκαταλείψουν τις, χω... τις περιοχές αυτές που έχουν καθυστερήσει. Έχουν πολλούς λόγους για τους οποίους έχουν καθυστερήσει. Δεν πρέπει να, ξεχάσουμε, να τους ξεχάσουμε και να τους αφήσουμε πίσω. Ένα, Ένα θέμα που είναι και το αγαπημένο μου Υπάρχει αναλφαβητισμός για τα θέματα του άνθρακα και ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης. Πρέπει να κάνουμε κάτι οπωσδήποτε. Για παράδειγμα, στα κτίρια πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι κτίριο χαμηλών εκπομπών ε, σε άνθρακα. Πρέπει νομίζω λοιπόν να αφιερώσουμε πάρα πολύ προσπάθεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Ελπίζω ότι η δική μου ε, περιοχή, που είναι μάλιστα πολύ ε, μεγάλη, θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιτύχει τους στόχους και πιστεύω ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα το λόγο. Ε, ποιος, ε, ποιος είναι εδώ, ο κύριος Παπαντονίου. Εντάξει, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύτιμη έκθεση της παρόλο που απουσιάζει. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα είναι πολύ χρήσιμα. Ιδίως στην πρακτική εξέταση των μέτρων για να πετύχουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα ή των μέτρων για να ξεπεράσουμε το 20%. Αυτό πραγματικά ήταν ένας από τους σκοπούς που θέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή μας θέλαμε να γίνει μια συζήτηση ε, συνειδητή για το όλο θέμα, στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, να δει και να δουν ποια είναι τα κόστη οι ωφέλειες και ποιο το κόστος ε, του να ξεπεράσουμε τα ποσοστά αυτά που έχουν τεθεί ως στόχοι για το 2020. Η έκθεση λοιπόν κάνει σχόλια εύστοχα, ιδίως σε σχέση με όσα υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον οδικό χάρτη της χαμηλής κατανάλωσης ε, του άνθρακα για τους μακροπρόθεσμους στόχους μας, για τη μείωση δηλαδή. Εδώ μιλώ για τις ιδέες σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να έχουμε τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και να είναι πιο αποτελεσματικές ώστε να έχουμε τρόπους περιορισμού των εκπομπών με φτηνά μέσα. Για την χρηματοδότηση και τα εργαλεία χρηματοδότησης, ο δικός χάρτης δίνει έμφαση και στην ανάγκη επενδύσεων εντό τη Ευρωπαϊκή οικονομίας, ιδίω στα κτίρια και τι μεταφορές. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και πώς επίση θα ευθυγραμμίσουμε την διτή αυτή προσέγγιση στο μέλλον και στα πλαίσια της δημοσιονομικής αναθεώρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό θα εξυπηρετήσει τις συζητήσει και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα επίκαιρη αυτή η έκθεση. Ελπίζουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί πριν δώσει τις ε, πρώτες της προτάσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την ενεργειακή αποδοτικότητα πραγματικά καλωσορίζουμε τα όσα προτείνονται, διότι και πάλι τονίζεται η σημασία αυτής της έννοιας. Πρέπει να τεθούν σχετικοί στόχοι και να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για να ξεπεράσουμε κάποια στιγμή το 20%. Επίσης, δύο πρόσθετες παρατηρήσεις. Νομίζω αρκετοί από τους ε, βουλευτές εδώ τα θύμισαν. Ε, ο στόχος των διεθνών διαπραγματεύσεων και της αντιμετώπισης των διεθνών προκλήσεων. Αυτό που θέλουμε όλοι να έχουμε κατά νου είναι ότι βρισκόμαστε σε διαφορετική θέση από ό,τι συνέβαινε πριν δύο ή τρία χρόνια, όταν μιλούσαμε για το ενεργειακό πακέτο. Τότε μιλούσαμε για μια μονομερή δέσμευση, ότι θα επιδιώξουμε το 20% και ότι θα εφαρμόσουμε την, την απαραίτητη νομοθεσία για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Τώρα ε, έχουν αλλάξει τα πράγματα γιατί εντωμεταξύ οι ηγέτες κατών κυβερνήσεων έχουν εκφραστεί υπέρ της ε, μείωσης και όλες οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν πλέον αναλάβει δεσμεύσεις, έχουν υποσχεθεί ότι θα ε, θα υλοποιήσουν συγκεκριμένε νομοθετικέ πράξει για να επιδιώξουν αυτού του στόχου. Έχουν αλλάξει λοιπόν τα, τα πράγματα μέσα στην τελευταία τριετία. Υπάρχει κίνηση σε διεθνέ επίπεδο. Βέβαια δεν αρκεί αυτό που έχει γίνει τώρα. Χρειαζόμαστε διεθνώ δεσμευτικέ ε, συμφωνίε και εάν σκεφτείτε το πενταετές κινέζικο πρόγραμμα όπως εγκρίθηκε θα καταλάβετε ότι η Κίνα μπορεί από το πρόγραμμα να περάσει πλέον κατευθείαν σε συγκεκριμένες δράσεις. Για τη διαρροή τώρα άνθρακα, κάτι που το επεσήμαναν αρκετοί βουλευτές, είναι ένα θέμα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Στο ενεργειακό πακέτο είχαμε αναλάβει κάποιες σημαντικές ε, πρωτοβουλίες για να περιορίσουμε τον κίνδυνο διαρροής του άνθρακα στις τεχνολογίες μεταφοράς ενέργειας. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα σύστημα συγκριτικής δειγματοληψίας για, την, για τον περιορισμό αυτού του φαινομένου και αυτό αποτέλεσε μέρος του συμβιβασμού που ενέκρινε πριν από δύο χρόνια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του ενεργειακού πακέτου. Τώρα, στον οδικό χάρτη και στις σχετικές συζητήσεις που κάναμε πρόσφατα εδώ, συνεχίζουμε τις προσπάθειες και παρακολουθούμε την κατάσταση. Σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, με το τι ίσχυε μάλλον πριν τρία χρόνια, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Γιατί και από την Κοπενχάγη έχουμε δει να εντείνονται προσπάθειες σε όλες τις χώρες, σε όλο τον κόσμο και επειδή η τιμή του άνθρακα τελικά είναι καλύτερη από αυτή που πριν, προβλέπαμε πριν από τρία χρόνια. Έχει φτάσει τα 20 ευρώ ανά κυβικό μέτρο διοξιδί του άνθρακα. Άρα τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι φανταζόμασταν. Φαίνεται λοιπόν ότι τα μέτρα που έχουμε προβλέψει είναι αποτελεσματικά, είναι εύστοχα και θα συνεχίσουμε να ε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Τότε η κυρία Καβάλιο θα απαντήσει και πάλι για την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα... Ε, ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα τα σχόλια τα οποία θα τα μεταφέρω στην κυρία Ρωμάν Τζόρνταν Σίσλεϊ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, βλέπουμε από τη συζήτηση, να λάβουμε υπόψη την καινοτόμο χρηματοδότηση, την πρόσφατη τεχνολογία και να επανεπενδύσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικές λοιπόν οι παρατηρήσεις που ε, έκαναν οι συνάδελφοι. Το βασικό θέμα όμως νομίζω ότι είναι η ευθύνη της ε, Επιτροπής μας να εξετάσει το ρόλο της ε, βιομηχανίας ε, σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών αερίων και του κινδύνου διαρροής άνθρακα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν διατάξεις, ε, χρήση για παράδειγμα του CDM και της ανακατανομής των ποσοστώσεων, όμως Πιστεύω ότι αυτές οι απόψεις βρίσκουν σύμφωνη την ε, συντάκτρια της γνωμοδότησης και η γενική άποψη του ΕΛΚ είναι ότι τα βασικά ζητήματα και η διεθνής ε, ε, συμφωνία έχει να κάνει ακριβώς με την επίλυση με, τη λύση για την βιομηχανία. Πρέπει να έχουμε καινοτόμε λύσεις που να λαμβάνουν υπο, υπόψη και να μπορέσουμε να προτείνουμε μία κάπως πιο ολιστική προσέγγιση, όπως κάνουμε ήδη στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, ε, για παράδειγμα, για τις ε, αεροπορικές μεταφορές. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να αποτελέσει μία προστιθέμενη αξία για τις ε, διεθνείς διαπραγματεύσεις, όπως επίσης και για τους ευρωπαϊκούς στόχους για τον διοξίδιο του άνθρακα. Κατά την άποψή μας, ε, η επόμενη συμφωνία δεν θα είναι απλή όπως ήταν αυτή του Κιώτο, θα είναι πολύ πιο περίπλοκη γιατί είναι πολύ πιο περίπλοκη η κατάσταση στον κόσμο. Δεν χρειάζεται απλώς να έχουμε δεσμευτικό στόχο, ε, πρέπει να έχουμε διαφορετικά σύνολα στόχων, ε, τομεακές συμφωνίες και θα μπορούσαμε από σήμερα να αρχίσουμε να αναλύουμε τις δυνατότητες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Θα μεταβιβάσω όλα σας τα σχόλια ε, στην κυρία Τζόρνταν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ για τις ε, τροπολογίες προθεσμία 21 Μαρτίου και μετά όπως ελέγχθη την Πέμπτη έχουμε το, την ακρόαση και όλοι είναι προσκεκλημένοι. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα και πρόκειται για την κοινή γεωργική πολιτική του 2020. Ο συνάδελφος Ρόντε είναι ο εισηγητής μας και είναι ο πρώτος και μοναδικός που θα λάβει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε, σχεδόν όλοι να συμφωνήσουμε, ότι η αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής χρειάζεται και επιγόντως. Ξέρω ότι είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Βρετανικής Προεδρίας στο ε, όταν θα έρθει η σειρά της. Οπότε ε, πρέπει να μπορούν οι γεωργοί να παράγουν ασφαλώς ε, τα προϊόντα τους σε ανταγωνιστικές τιμές για τους γεωργούς και εάν έχουμε μία σωστή πολιτική για την πράσινη ενέργεια θα είναι προς όφελος όλων πρόκειται ε, για έναν πόρο που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί στη Γεωργία, δηλαδή οι Γεωργοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να υποφεληθούν αυτού, αυτής της δυνατότητας και θέλουμε να έχουν τη δυνατότητα να ε, ε, επενδύσουν ή στις βιώσιμες μεθόδους Βέβαια εδώ δεν αναφερόμαστε στην περιβαλλοντολογική πτυχή. Ε, ε, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την ε, πράσινη διάσταση. Θέλουμε να μπορέσουν οι γεωργοί να έχουν την δυνατότητα απασχόλησης σε άλλες δραστηριότητες που δεν είναι αμυγός διεθνής γεωργικές και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο απλό, διαφανή και για τους ε, γεωργούς και για το κοινό. Οπότε ε, εάν ε, υπάρχουν τρία από τα δέκα δημόσια αγαθά νομίζω ότι θα είναι προς όφελος των γεωργών. Τα σημεία όμως εκκίνησης διαφέρουν αναλόγως των κρατών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε όλοι οι γεωργοί να έχουν τις ίδιες δυνατότητες στην υποδοχή των οικολογικών συντελεστών, δηλαδή όλες οι παράμετροι να ληφθούν υπόψη, διότι πιστεύω ότι ο οικολογικός συντελεστής θα είναι προς όφελος του περιβάλλοντος, θα δώσει δυνατότητες ανάπτυξης στους γεωργούς και θα αυξήσει τη διεθνή ε, ανταγωνιστικότητα ανταγωνιστικότητά μας. Ε, ε, προσβλέπω στα σχόλια των Επιτροπών και θα συνεργαστώ με τους σχιώδεις εισηγητές για να μπορέσουμε να έχουμε μια ισχυρή πρόταση για το μέλλον της κοινή γεωργικής ε, πολιτικής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πυλό είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η γεωργία παραμένει ένας τομέας ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει πολύ σημαντικά σε ΑΕΠ και σε άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Η στρατηγική του 2020 έχει αναθέσει στην ΚΑΠ τον ρόλο του θεματοφύλακα της επισητιστικής ασφάλειας και της παραγωγής τροφίμων. Επίσης παράγοντα πρόθεσης της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και της διαφοροποίησης του 8ου προγράμματος πλαισίου, της έρευνας που θα προκύψει δηλαδή από τις νέες αυτές ευκαιρίες. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συζήτηση που γίνεται σήμερα και τον ιδιαίτερο ρόλο που αποδίδει στην γεωργία, την περιβαλλοντική προστασία και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Οι προτάσει του εισηγητή Ρόντε είναι συστάσει που μπορούμε να τι συμμεριστούμε. Αλλά θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνολογική διάσταση τη γεωργία, καθώ και την δυνατότητά τη να παρέχει πράσινη ενέργεια, οικολογική ενέργεια καθώς και όπως λέει παράγραφος 5 να συμπεριληφθεί το στοιχείο αυτό στον πρώτο πυλώνα. Επίσης για την ε, μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κονδύλια πριν ε, σε ένα πλαίσιο πολιετές αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι πρακτικές που έχουν ιστορική πορεία μακρά μπορεί να αποτελούν και πολιτιστικό αλλά και περιβαλλοντικό κληροδότημα. Να σκεφτούμε επίσης αγροτικοπεριβαλλοντικά μέτρα για να δημιουργηθούν τέτοια προϊόντα που διατομεακά και στον πρώτο και στον δεύτερο πυλώνα να, ε, να προστατεύονται. Να υπάρχει μάλιστα πρόσβαση σε μέτρα για την βιωσιμότητα, την πιστοποίηση και την τεχνολογική στήριξη. Η παγκοσμιοποίηση έχει ε, επιδεινώσει την, ε, το ευάλωτο των ε, επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη, καθώς η πρόσφατη κρίση έχει πλήξει όλους τους τομείς της γεωργικής παραγωγής και δείχνει πόσο πρέπει να προστατευτεί η σημερινή ΚΑΠ. Τα μέτρα μας δεν είναι αρκετά ευέλικτα θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη και ακραίε καταστάσει διακύμανση των τιμών. Αυτό το θεωρώ κρίσιμη σημασία και θα πρέπει να το σκεφτούμε στα πλαίσια τη αναθεώρηση τη ΚΑΠ. Να έχουμε μέτρα για την καταπολέμηση των οικονομικών κύκλων και να συμπεριληφθούν στον πρώτο πυλώνα, ώστε να μπορεί η ΚΑΠ να ανταποκριθεί αυτομάτω και εγκαίρω στι ε, διακυμάνσει τη αγορά. Επειδή υπάρχουν φυσικέ καταστροφέ που δυστυχώ ολοένα και παραλαμβάνονται συχνότερα τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά δείχνουν ότι το, κερδοφορία των γεωργικών επιχειρήσεων συνεχώς απειλείται. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε ε, τρόπους παρέμβασης πιο αποτελεσματικούς και να προστατεύσουμε επίση το εισόδημα των γεωργών. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε κριτήρια πιο ισότιμα, πιο δίκαια, ώστε να ληφθεί υπόψη το πραγματικό κέρδος και το κόστος ζωή των γεωργών στι διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. καθώς και σε σχέση με τη διακύμανση της ίδιας τους της παραγωγής. Ω προ την ανάπτυξη του υπαίθρου πρέπει να ε, ενισχυθεί ο δεύτερο πυλώνα ώστε να υπάρχουν και μέτρα επένδυση για επιχειρήσει που προτιμούν την βιώσιμη γεωργία και την υποστηρίζουν. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό ε, πακέτο και για τους νέους όταν ξεκινούν για πρώτη φορά τις γεωργικές τους δραστηριότητες να τους προτείνουμε ενημέρωση, πρόσβαση στη γη ε, και δυνατότητα εκπαίδευσης για να γίνουν πολυαποτελεσματικέ οι επιχειρήσει του. Να παρασκευθούν οι απαραίτητε υπηρεσίε επίση και να καλυφθούν οι ανάγκε όσων παραμένουν στι περιοχέ τη υπαίθρου. Ω προ τον πληθυσμό ακριβώ τη υπαίθρου, στι ε, ορεινέ περιοχέ, εκεί θα πρέπει να προβλεφθεί και πρόσβαση ε, σε γεωλογικούς ε, πόρους προκειμένου να προληφθεί και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Εδώ λοιπόν θέλουμε να περάσουμε σε μια εξυγχρονισμένη ευρωπαϊκή γεωργία. Εύχομαι λοιπόν στο μέλλον οι διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει για την ΚΑΠ να οδηγήσει στο διάστημα 2014-2020 στην δημοσιονομική κάλυψη του γεωργικού κλάδου που είναι τόσο καθοριστικός για την ευρωστία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κρίτς. Ξέρω ότι έχετε μεγάλες δυσκολίες να προφέρετε το όνομά μου. Σκρουμπζουπ. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ευχαριστώ. Όντως, Υπάρχουν ε, τρεις ε, απόψεις εδώ. Δηλαδή, αφενός υπάρχει η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέχρι το 2020 και πρέπει να ε, ανταποκριθούμε στις προκλήσεις όσον αφορά τη διατροφή και τα τρόφιμα και εδώ αναφερόμαστε και στη συνοχή. Όχι μόνο τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μελών και των περιφερειών διότι η Ήπεθρος εκπροσωπεί το 98% της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρα ε, αν νομίζουμε ότι είναι ένα επουσιώδες θέμα νομίζω ότι πρόκειται για μεγάλη πλάνη. Δεύτερον ε, θέλω να, ε, να απαντήσω εις την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει της οποίας καταρτήσαμε μία έκθεση η οποία θα πρέπει ούτως ή άλλως να, ε, ε, ε, να αντιμετωπίζεται στην έκθεση του κυρίου Ρόντε διότι η συμφωνία υπάρχει στα πέντε σημεία όχι στα οκτώ διότι τα άλλα τρία αναφέρονται σε άλλες πτυχές της γεωργικής πολιτικής και πρέπει να σας πω ότι οι θετικές μου, τα θετικά μου σχόλια, ποια είναι τα θετικά μου σχόλια στην έκθεση Ρόντε όπου λέγει ότι θα πρέπει ο οικολογικός συντελεστής να περιοριστεί στον πρώτο πυλώνα. Αυτό συνάδει με την ανακοίνωση, αλλά υπάρχει συγγητή σε άλλη επιτροπή που συνιστά να τοποθετηθεί ο οικολογικός συντελεστής στο δεύτερο πυλώνα. Και ο εισηγητής άλλωστε εδώ μιλά και λέει ότι ο οικολογικός συντελεστής δεν χρειάζεται να αυξηθεί τώρα. Εγώ όμως αμφιβάλλω σχετικά με αυτή τη δήλωση διότι πιστεύω ότι πρέπει να επιλέξουμε ε, τρεις ε, ε, τρεις συντελεστές από δέκα. Πουθενά όμως δεν είδα να αναγράφεται ότι υπάρχουν 10 απαιτήσει. Η Γεωργική Επιτροπή, η Επιτροπή Γεωργίας αναφέρεται σε 11 αλλά ε, υπάρχουν και θέματα σχετικά με τα ζώα. Ε, τα υπόλοιπα όμως ε, δεν πρέπει να τα παραβλέψουμε όταν μιλάμε για οικολογικούς συντελεστές. Είναι κάτι λοιπόν που πρέπει να μας απασχολήσει, όπως επίσης πρέπει να αναρωτηθούμε αν χρειάζονται τρεις ή όπως λέγει η Επιτροπή Γεωργίας δύο οικολογικοί συντελεστές στους οποίους πρέπει να συμμορφωθούν οι γεωργοί για να διαχειριστούν τις πληρωμές. Ε, εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η γεωργία έχει και αυτή την άλλη οπτική γωνία, δηλαδή εκτός της παραγωγής παράγει γενικώς αγαθά και ο οικολογικός συντελεστής αναφέρεται στην ε, πολιτική γεωργίας μέχρι το 2020 και πρέπει να πούμε ότι η γεωργία στην Ήπεθρο ε, ε, παράγει ορισμένα δημόσια αγαθά τα οποία διατίθενται δημόσια. Άρα και αυτό είναι οικολογικό και επίσης ε, ε, δεν περιορίζεται εις ε, τα διατροφικά αγαθά και στην ενέργεια η παραγωγή της γεωργίας αλλά επηρεάζει και την ανάπτυξη της βιομηχανίας του εμπορίου και άλλων τομέων της οικονομίας. Πρέπει λοιπόν να σταθμίσουμε τις συνέργειες μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και των άλλων πολιτικών που δημιουργούνται και αυτό συνάδει με τους στόχους της στρατηγικής για το 2020. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε το, τις συνέργειες οι οποίες δημιουργούνται σε περίπτωση που οι πολιτικές ε, εφαρμοστούν σωστά. Άλλωστε, υπάρχει και δημιουργία ποιών ενεργείας, όχι μόνο ανανεωσίμων, αλλά ένα κλασικό θέμα εδώ είναι η αναθεώρηση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής στον τομέα της ζάχαρης. Έχουμε ε, ε, χάσει ήδη 16.000 θέσεις εργασίας με την αναθεώρηση της πολιτικής και την κατάργηση της καλλιέργειας ζαχαροτέφλων και ε, υπάρχουν και πολλά αγροκτήματα στην Ευρώπη που πρέπει να αποτελέσουν τον πρώτο στόχο μας, δηλαδή να δημιουργηθούν εκεί θέσεις εργασίας και παραγωγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλά ε, προϊόντα νέα, πολλές εφαρμογές νέες και η καινοτόμα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εφαρμόσει μεθόδους καινοτόμες όχι μόνο στην παραγωγή και στην ενέργεια αλλά και σε άλλους τομείς. Και ε, καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι πέραν των άλλων στόχων ο στρατηγικός ρόλος του περιβάλλοντας πρέπει επίσης να τονιστεί διότι βλέπετε ότι σε πολλές περιοχές του κόσμου υπάρχουν αναταραχές που αναφέρονται στην αύξηση των ε, τιμών τροφίμων και η Ευρώπη εδώ εμπλέκεται γιατί εισάγουμε 70% του εξαγωγικού μας εμπορίου από υποανάπτυξη χώρες. Η Γεωργία λοιπόν μπορεί ε, να είναι μια πηγή πόρων ε, πιο σημαντική από ό,τι στο παρελθόν για την ενέργεια αλλά πέραν αυτού και για άλλους τομείς και για να δημιουργηθούν αυτές, ε, αυτοί οι πόροι δημιουργούνται και εκπομπές και αυτό είναι αρνητικό. Μέχρι στιγμής λοιπόν πρέπει να πούμε ότι έχουμε αποδώσει μεγάλη σημασία εις ε, τα δάση για να μειωθούν οι εκπομπές χωρίς να αναφέρουμε τον ρόλο που μπορεί να παίξει η γεωργία στον τομέα αυτό με ε, την ε, αφομοίωση των οργανικών ουσιών του εδάφους και περιορίζοντας την διαδικασία οξυδωσης και ε, των, ε, των συστατικών που βρίσκονται στο έδαφος. Λοιπόν, με μία αύξηση 0,5% αυτών των παραμέτρων μπορούμε να μειώσουμε πολύ το διοξίδιο του άνθρακα και εδώ πρέπει να αναφερθούμε σε ορισμένα βασικά θέματα. Και Γι' αυτό θα έλεγα ότι η γεωργία μπορεί να προκαλέσει ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και ε, να ε, χρησιμοποιήσουμε ε, διασυνδέσεις και προς άλλες βιομηχανίες, ε, την αυτοκινητοβιομηχανία παραδείγματος χάρη και να ε, μπορέσουμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα της ενέργειας των οχημάτων δηλαδή θα βοηθηθούμε πολλαπλώς με μια ενεργειακή βελτίωση ε, ε, βελτίωση και της ενέργειας θερμότητος διότι ναι μεν καταναλώνουμε ενέργεια για την ψήξη αλλά μπορούμε και να επανακτήσουμε ενέργεια από αυτή την πηγή βέβαια το θέμα είναι σε τι, με τι κόστος οπότε εάν ήταν δυνατόν θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας και την ε, ε, τον δεύτερο πυλώνα και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στον ε, τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μία καλύτερη υποδομή, με καλύτερη διασύνδεση μέσω του ευρυζωνικού διαδικτύου και με στοιχεία τα οποία είναι υπέρ της ε, μειώσεως ε, των εκπομπών, αυξάνοντας την ηλιακή ενέργεια ή ε, ανακτώντας την ενέργεια που δαπανάται ή την ύπεθρο για την ψήξη ή ε, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτηρίων. Αυτά είναι τα σχόλια που ήθελα να παρουσιάσω και ε, θα συνεργαστώ με τον εισηγητή για τη διατύπωση προτάσεων που δεν θα ε, καταστρέψουν την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης αλλά θα μπορέσουν να μας δώσουν τη δυνατότητα να τονίσουμε καλύτερα το ρόλο του τομέα αυτού ο οποίος ε, συνάδει με τους στόχους της Επιτροπής μας. Η κυρία Εκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο ρόλος μας ε, ως Επιτροπής Βιομηχανίας ε, Έρευνας και Καινοτομίας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει να ε, δούμε τους γεωργούς και τους επιχειρηματίες όπως πραγματικά είναι και πρέπει να δούμε και ε, τι γίνεται με τις θέσεις απασχόλησης και στον τομέα της γεωργίας αλλά και της δασοκομείας. Ε, θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες είναι σημαντικές στο κείμενο της Ήτρε και για παράδειγμα πρόκειται για το ρόλο της βιομηχανίας και των θέσεων απασχόλησης, όπως επίσης και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και αν δούμε, ας πούμε, την πράσινη διάσταση, το πράσινο στοιχείο θα πρέπει να είναι στο πρώτο πυλώνα. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν ευκολότερο και στα κράτη-μέλη θα σήμαινε ένα σύνολο αρμοδίων αρχών, ενώ στο δεύτερο πυλώνα υπάρχουν διάφορες κυβερνητικές ε, ε, υπηρεσίες ε, και γραφεία που υπησέρχονται, οπότε για μένα ο πρώτος πυλώνας είναι καλύτερος και ειδικότερα αν θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε τον τομέα ώστε να είναι πιο σύγχρονος και πιο ανταγωνιστικός, νομίζω ότι στον πρώτο πυλώνα μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Είναι πραγματικά τραγικό να βλέπουμε την ε, κρίση, την ε, τρέχουσα, το κλίμα ε, και η ενέργεια έχουν δημιουργήσει ακόμη χειρότερα προβλήματα. Βλέπουμε τι έγινε και στην Ιαπωνία που θα προσθέσει ακόμη μεγαλύτερο βάρος σε όλη αυτή τη διαδικασία οι δυνατότητες χρήσης αποβλήτων από ε, γεωργική παραγωγή για την δημιουργία βιολογικού αερίου είναι πάρα πολύ σημαντική και για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας ε, ε, και και για τους λόγους που ανέφερα υπάρχουν οι δυνατότητες αλλά δεν υπάρχουν οι επενδύσεις και νομίζω ότι η Γερμανία είναι ένα παράδειγμα μπορούμε να δούμε δηλαδή τέτοιου είδους δυνατότητες στη Γερμανία, Αλλιώ πρέπει να ε, δούμε την περίπτωση της Νέας Ζηλανδίας για παράδειγμα. Πρέπει να υπάρχουν κινήτρα για τους γεωργούς να επενδύσουν στη γεωργική παραγωγή και πιστεύω ότι αν δούμε το υλικό ε, της Επιτροπής Γεωργίας αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα για την αχρανάπαυση και βλέπουμε τις ανάγκες ε, για κάψιμα και για τρόφιμα στο μέλλον, στο μέλλον νομίζω ότι είναι τρομερό να έχουμε 5% ε, κριτήριο για αγρανάπαυση. Νομίζω ότι από περιβαλλοντική απόψης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το, τη γη μας και ίσως θα έπρεπε ε, να χρησιμοποιήσουμε τα απόβλητα για, να, για την παραγωγή ε, βιολογικού αερίου. Ε, ακόμη και ε, οι, κοινων, οι κοινωνικοί μας εταίροι μας λένε μην χρησιμοποιείτε αυτό το 5% χρειαζόμαστε τη γη για να παράγουμε τρόφιμα, προϊόντα και καύσιμα. Λοιπόν, το 5% της αγρανάπαυσης σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ παροχημένος τρόπος για τη βελτίωση της γης μας και της βιομηχανίας, όπως επίσης και την παραγωγή από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο χρησιμοποιήσαμε, ε, το οποίο, οποίο αναφερθήκαμε σήμερα το πρωί, για πολλά άλλα ζητήματα και ισχύει και για τη γεωργία. Υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια που αναφέρουν τις δυνατότητες που υπάρχουν για, για ενεργειακή αποδοτικότητα ε, με, ε, σε ποσοστά 40 με 50%. Δεν υπάρχει δυνατότητα στο πλαίσιο της ΚΑΠ να το επιτύχουμε αυτό, αλλά σε τομέα της απασχόλησης είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, η νέα ΚΑΠ να έχει τέτοιου είδου εργαλεία. Ευχαριστώ. So, dann darf ich noch der Kommission das Wort geben. Δώσω ακόμη το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θα αναλάβει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς ε, την Επιτροπή σας ε, για την ε, σημασία που δίνει στην ανακοίνωση για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς βλέπω ότι θετική προσέγγιση στις προτάσεις που αφορούν την πράσινη διάσταση Νομίζω ότι είναι ε, μία προσέγγιση που ε, μοιάζει αρκετά με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η έκθεση, όπως και κάποιοι από εσά επέμειναν στην αναγκαιότητα αυτή η πράσινη διάσταση να μην σημαίνει επιπλέον γραφειοκρατία. Και αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερος Γνωρίζετε ότι η ΚΑΠ έχει ε, υπάρξει αντικείμενο απλοποιήσεων ε, και ειδικότερα μέσω της ανακοίνωσης αυτής. Για παράδειγμα, υπάρχει μια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ε, για να εξασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες πληρωμών, γεωργικών πληρωμών ε, αλλά και ε, οι εκπρόσωποι των γεωργών ε, συμμετέχουν και επαγρυπνούν προκειμένου τα μέτρα αυτά να μην επιφέρουν επιπρόσθετη γραφειοκρατία. Αντιθέτως, να οδηγηθούμε σε λιγότερη γραφειοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί επίσης ε, απολύτως με την άποψη την, ε, επί της Επιτροπής ε, για τη σημασία της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων λύσεων για τη γεωργία. Στην ανακοίνωση συγκεκριμένα όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σαφής ότι το περιβάλλον, η κλιματική μεταβολή η καινοτομία στο τομέα της γεωργίας είναι αρχές ε, οι οποίες θα αποτελούν τμήμα των προσεγγίσεων και των μέτρων ε, που θα ε, εφαρμοστούν για την ανάπτυξη της υπέδρου, Στο πλαίσιο της καινοτομίας πρόκειται να εκπονηθεί μια, ένα έγγραφο συγκεκριμένα για την καινοτομία στον τομέα των, ε, ε, της γεωργικής παραγωγής, ε, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και παράδειγμα της κλιματικής μεταβολής, με σκοπό την αύξηση ή τη διατήρηση της παραγωγής, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους και με σκοπό την βελτίωση της ε, γεωργικής πολιτικής ε, λαμβάνοντας υπόψη ε, την διαχείριση των υφισταμένων πόρων. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ρόντε έχει πάλι τον λόγο και θα ήθελα εδώ να απαντήσω. Δανικά, δανέζικα και παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ήταν όλα επικοδομητικά. Νομίζω ότι από αυτής της βάσης μπορούμε να διπραγματευτούμε εάν θέλουμε να καταρτήσουμε μια πλήρη έκθεση για αυτό το θέμα. Εδώ λοιπόν, ε, στα πλαίσια μιας τέτοιας περιορισμένης γνωμοδότησης, με τους 115 χαρακτήρες που επιτρέπονται, είναι με τους 1500 χαρακτήρες που επιτρέπονται, είναι αδύνατο να τα καλύψουμε όλα. Όμως, θέλω να διαμορφωθεί ένα σχέδιο γνωμοδότησης που να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των παρατηρήσεων που έγιναν. Er øh, Βεβαίω, ε, για το έγγραφο αυτό να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια γενική γνωμοδότηση. Ε, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση σε στοιχεία σημαντικά, ώστε η γεωργία να παραμείνει ένας τομέας στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας. Όπως είπε η κυρία Εκ, θα πρέπει να γίνει μια πραγματική επιχείρηση η γεωργία για να συνεισφέρει μαζί με, τις υπόλοιπες, ε, με τα υπόλοιπα εγχειρήματά μας ε, στην, στους στόχους της στρατηγικής το 2020. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε το περιθώριο λιγμών που διαθέτουμε ακόμα και πριν την υποβολή των τροπολογιών και να σκεφτούμε ότι η έκθεση μπορεί να γίνει πολύ πιο μακροσκελής αν γεμίσει από πάρα πολλές τροπολογίες. Αλλά παρόλα αυτά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μια έκθεση αδιάσυστη σημασίας. θα πρέπει και οι υπόλοιπες επιτροπές να μπορούν να διαβάσουν την γνωμοδότησή μας και κάνω έκκληση προς τους συναδέλφους να ενημερώσουν για όλα αυτά γιατί υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες από τον οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Er θα μπορούσαμε λοιπόν για τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα να διαπραγματευτούμε διότι στον πρώτο πυλώνα ό,τι μεταφερθεί ε, σαφώς ε, έχει να κάνει με τα κίνητρα που μπορεί να δοθούν προς την γεωργία. Και σας ευχαριστώ για τα ιδιαίτερα σχόλια και τα επικοδομητικά σχόλια που κάνετε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. 22 Μαρτίου 12 το μεσημέρι είναι η λήξη της προθεσμίας για κατάθεση τροπολογιών και τώρα έρχομαι στο επόμενο θέμα ε, που αναφέρεται ε, εις ε, στο θέμα που θα παρουσιάσει η συνάδελφος Φόρντ και πρέπει να δούμε ε, αντιμέτωπη δηλαδή στο πρόβλημα της ασφαλείας των υπερακτήων δραστηριοτήτων με εκμετάλλευση συντασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και θα διαθέσουμε μισή ώρα στη συζήτηση αυτή. Η κυρία Φόρντ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε για το θέμα. Είχαμε μια συνάντηση με τους εισηγητές την περασμένη εβδομάδα και συνέταξα μια έκθεση που νομίζω ότι έχει μοιραστεί σε όλα τα μέλη. Εδώ λοιπόν υπήρχε αυστηρό όριο για τους χαρακτήρες, οπότε πολύ περισσότερο θα θέλω να είχα συμπεριλάβει, αλλά νομίζω ότι είναι και πολλά αυτά που θα συμφωνήσουμε με τους ε, συγητές για τις τροπολογίες, οπότε θα καλύψουμε πολλά. Στα πρώτα όλα στάδια κοιτάζαμε τις ε, περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχουν περισσότερες υπεράκτιες δυνατότητες, κάποια που μπορούν να ελιμενιστούν, οι νέε περιοχές που αρχίζουν να θεωρούνται υπεράκτιε. Εδώ επικεντρωνόμαστε στο πετρέλαιο βεβαίως και τις ανάγκες μας σε φυσικό αέριο. Για τον, για τον κόλπο του Μεξικού λοιπόν και τα όσα εκεί μας απασχόλησαν θα πρέπει να σκεφτούμε και τις τιμές και την ασφάλεια στα δικά μας τα ύδατα και βεβαίω προ όφελο όλων μας θα είναι ως προς την ενεργειακή ασφάλεια και την διαφοροποίηση της προμήθειας να διατηρήσουμε την εγχώρια προμήθεια για να είμαστε ασφαλείς. Θα ήθελα οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στόχο να έχει να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα ύδατα και να μην υπονομεύσει τις ισχύουσες προδιαγραφές. Να αποφύγουμε την γενίκευση διότι η εξόριξη είναι ένα θέμα, επίσης υπάρχουν μεγάλες πιέσεις εδώ, υπάρχουν ε, πηγάδια τα οποία λειτουργούν με χαμηλότερη πίεση, με υψηλότερη. Θα πρέπει λοιπόν η κάθε περιοχή και το, η κάθε περίπτωση να εξετάζεται με βάση τον δικό της ε, συγκεκριμένο κίνδυνο. Στη Βόρεια Θάλασσα Λόγου χάρη, είδαμε οι Αμερικανοί να έχουν ε, ένα, μια προσέγγιση tech box, όπως θα μπορούσαμε να την πούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως επεσήμανε διάφορα θέματα ασφαλείας. Θα πρέπει διαρκώς λοιπόν για σκοπούς ασφαλείας να κάνουμε αξιολόγηση των κινδύνων, να βλέπουμε τους περιβαλλοντικές και τεχνικές απαιτήσει τα ζητήματα αυτά για κάθε περίπτωση εγκατάστασης, για κάθε συγκεκριμένη υπόθεση να τα εξετάζουμε προσεκτικά. Θα πρέπει έτσι να υποχρεώνουμε τους ε, φορείς και τους ε, υπευθύνους των εταιριών να αξιολογούν πλήρως όλους τους κινδύνους εκ των προτέρων που ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία και δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι σωστά έχει ορίσει τα θέματα της ασφάλειας, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά τα κριτήρια ασφάλειας από τους δύο φορείς και ανεξάρτητους έλεγκτες και να δούμε ότι κάποιες φορές οι φορείς κάνουν αλλαγές στις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ε, αυτό δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Θα πρέπει να ακολουθείτε αυστηρό το καθεστώ βέλτιστων πρακτικών και το σύστημα βέλτιστων πρακτικών όπω ισχύει σε κάποια ευρωπαϊκά κράτα. κράτη. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχει ένα ιστορικό για τι προδιαγραφέ ε, υγεία και ασφάλεια όπω και στον γεωργικό τομέα. Πολύ καλό είναι αυτό η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων να λαμβάνεται υπόψη, όχι μόνο η ασφάλεια των προϊόντων. Όμως οι διαδικασίες ασφαλείας είναι εξίσου σημαντικές και να σας εξηγήσω ότι εννοώ. Στην περίπτωση του ΡΕΓ φαινόταν ότι οι βασικές διαδικασίες για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαζομένων ε, είχαν ακολουθηθεί. όμως δεν είχε δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν είχαν γίνει δοκιμές δεν υπήρχαν αυτόματα, ή μάλλον οι αυτόματες διαδικασίες πάυσης λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος Δεν ε, εφαρμόστηκε πλήρωση Το είχαν παρακάμψει παρά τις βέλτιστες πρακτικές Και υπήρχε μεγάλη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί πριν πατήσουν το κουμπί του συναγερμού σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα έχει επιτρέψει το ρυθμιστικό καθεστώς. Θα πρέπει αυτά να τα δούμε σε σύγκριση με τόσα συμβαίνουν σε είδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και κάπως πιο όρημα από την πλευρά της αντιμετώπισης των αρχών. Να σκεφτούμε λοιπόν και την ασφάλεια των διαδικασιών και της ε, εκπαίδευσης των εργαζομένων. Είναι σημαντικά τα θέματα αυτά, αλλά εξίσου σημαντική, όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι και η υλοποίηση, η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας από εξόριξη στη θάλασσα θα μπορεί να συγκριθεί μόνο με το πόσο αποτελεσματικοί είναι οι ελεγκτές και οι νομοθέτες. Η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων σε ορισμένα σημεία της ε, Μεσογείου ή της Μαύρης Θάλασσας είναι σημαντικό, δίνει ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες προσπάθειες. Οι ελεγκτές θα πρέπει να συνεργάζονται με τους φορείς απευθείας και να έχουν επαρκή ενημέρωση και γνώσεις για να μπορούν να αξιολογούν τις μεθόδους εργασίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αφώς ο ελεγκτής που χρησιμοποιήθηκε ήταν ε, ε, ε, ανεπαρκής. Επίσης το οικονομικό καθεστώς θα πρέπει να είναι Η βιομηχανία να πληρώνει τα κράτη-μέλη να μπορούν να αξιοποιήσουν μάλιστα τα κονδύλια αυτά. Και εάν υπάρχουν περιορισμένοι πόροι για την εξέβρεση ελεγκτών με την απαραίτητη πείρα και εμπειρογνωμοσύνη, καθώς ήδη υπάρχουν ζητήματα πρόσληψης ακόμη και σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχει πιο προηγμένη βιομηχανία, θα πρέπει παρόλα αυτά αυτή η δυνατότητα να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Δεν είμαι επιπισμένη ότι θα είναι επωφελής μια απολύτως ε, νέα αρχή ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, εδώ μπορεί να έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει η κάθε ευρωπαϊκή χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδράμει. Δημιουργώντας νέες θέσεις σε τελείως νέους τομείς. Για διασυνοριακούς λόγου χάρη ερεγκτές, εφόσον μιλάμε για εγκαταστάσεις που βρίσκονται μεταξύ δύο κρατών. Επίσης πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών νομίζω ότι μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα και από την ΕΜΣΑ για να υπάρξει συντονισμός των όλων προσπαθειών. Αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει στη Βόρεια Θάλασσα, λόγου χάρη, είναι ο συστηματικός διάλογος μεταξύ των ελεγκτών. Έτσι λένε. Συναντιούνται συστηματικά, υπάρχουν ε, τέτοια ραντεβού και συμμετέχουν και μη ευρωπαϊκέ χώρε όπω η Νορβηγία που συμμετέχει σε αυτό το φόρουμ για τη θάλασσα. Νομίζω κάτι ανάλογο θα μπορούσε να γίνει και αλλού. Θα ήταν εξίσου εξυπηρετικό όπω στην Μεσόγειο. Στην Μεσόγειο. Στο ΜΕΝΤ, διότι η εξόριξη που γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει δεν γίνεται αναγκαστικά σε ευρωπαϊκά ύδατα. Το να συμμετέχουν λοιπόν στι ζητήσει, μη ευρωπαίοι εταίροι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης νομίζω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών βοηθά και στην καλύτερη κατάρτιση διεθνών προδιαγραφών. Η ασφάλεια και η ιδιοκτησία είναι δύο θέματα που αναπτύσσει εντατικά η έκθεση. Δεν είμαι όμω βέβαιη ότι για την ώρα έχουμε επαρκή στοιχεία. Τα κράτη, οι συμβουλευτέ μάλλον, θα πρέπει να σκεφτούν κατά πόσον στοιχεία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν όπως η αεροπλοεία που θα παρακολουθεί τα διάφορα συμβάντα για την πετρελαϊκή εξόρυξη και θα τα ε, επισημαίνει. Ή οποιοδήποτε μέσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την βελτίωση των διεθνών προδιαγραφών και το πώς λειτουργούν οι ελεγκτές και το πώς γίνεται η παρακολούθηση. Χρειαζόνται επίσης περισσότερα προγράμματα για την αντιμετώπιση κατεπηγόντων περιστατικών από τα βαθύτερα ύδατα λόγου χάρη και εφόσον υπάρχουν περιστατικά εκεί στην εξόριξη θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα πιο ταχύ. Ήδη στη Βόρειο Θάλασσα προβλέπεται να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα το οποίο θα το καλύψει οικονομικά η βιομηχανία και θα θέλαμε τέτοια συστήματα να διατεθούν σε όλε τι θαλάσσιε λεκάνε τη Μεσογείου, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν σκεφτούμε όμω πόσα πράγματα γίνονται ταυτόχρονα, το ΜΕΝΤ χάρη, το θέμα τίθεται ποιο θα τα πληρώσει, ποιο θα τα καλύψει. Στην Βόρεια Αφρική, εάν εμεί θα καλύψουμε το κόστο και το καθεξή. Ο εξοπλισμό ε, για την προστασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να είναι κατάλληλος για, διάφορες για διάφορα περιστατικά. Στον κόλπο του Μεξικόλογου χάρη είχαν χρησιμοποιηθεί εργαλεία τέτοια που να μπορούν να περιορίσουν την κοιλίδα. Τέτοια θα θέλαμε να διατεθούν και στις περιπτώσεις εξόρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως στη Βόρειο Θάλασσα και την Μεσόγειο. Εδώ τώρα υπάρχει και η αρχή ο πληρώνει και αυτή πρέπει να την έχουμε υπόψη, διότι οι μικρότεροι φορείς στην αγορά δεν μπορεί να επιβαρύνονται περισσότερο από τους μεγάλους και χρειάζεται συντονισμός των συμβασιούχων με τους φορείς και τα κονδύλια που πηγαίνουν προς τη βορειοανατολική θάλασσα από την Δανία και προς τις Φερόες είναι σημαντικά στοιχεία. Οι ΜΕΝ αντισταθμίζουν την ρήπανση των ΔΕ με 20 εκατομμύρια δολάρια ένα περιστατικό. Αυτή η εξοδετερώση του κινδύνου οδηγεί σε έναν βαθμό αυτοελέγχου των φορέων. Κοιτάζουν εκείνοι αν οι γείτονέ του σέβονται τι προδιαγραφέ. Ένα τέτοιο κονδύλι, ένα τέτοιο ταμείο θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να χρησιμοποιηθεί και σε άλλε περιπτώσει ευρωπαϊκών υδάτων. Θα πρέπει επίση να τεθεί ένα ανώτερο όριο. Εάν κανεί περάσει τα 250 λόγου χάρη, να συνεχίζει να είναι υπόλογο ο φορέα, αλλά αμέσω να προβλέπεται και μία. Ε, ένας μηχανισμός για την κάλυψη των ενοχικών υποχρεώσεων. Επίσης, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πιστεύω θα πρέπει να υποχρεώνονται να εφαρμόζουν τις προδιαγραφές ε, για τους ίδιους τους φορείς τους και Χρειάζεται εδώ μια πρακτική λύση για τον συνδυασμό των διαφορών ρυθμιστικών συστημάτων. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν εθνικοί ελεγκτές, αλλά θα ταξιδεύουν εκείνοι σε όλο τον κόσμο, θα ελέγχουν πώς λειτουργούν οι εξορίξεις σε όλες τις ε, περιπτώσεις. Ε, οι μέτοχοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τις βέλτιστες, πρακτικέ πρακτικές ε, ανά τον κόσμο. Σε γενικές γραμμές αυτός είναι ο σκελετός της συλλογιστικής μου. Ε, το αέριο, η έμσα, αυτά είναι πράγματα που θα προσθεθούν και με μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ με τους συναδέλφους για τις περιπτώσεις του ΜΕΔ και της Μαύρης Θάλασσας. Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις προσπάθειες αυτές τις περιοχές και να δούμε πώς θα συνδυάσουμε την ε, ε, δράση όλων των χωρών που έχουν σύνορα κοινά εντό ευρωπαϊκών υδάτων και εκτός. Γιατί ό,τι συμβαίνει εκτός μπορεί παρόλα αυτά να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, 29 Μαρτίου η ομάδα μου θα οργανώσει ακρόαση οι, οι σκεώδεις πρότειναν να έχουμε συγκεκριμένου προσκεκλημένους, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι επίσης. Θα έχουμε μιλητές από τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Θάλασσα, που ξέρουν από πρώτο χέρι τι έγινε στον κόλπο του Μεξικού και περιμένουμε απλώς κάποιες ε, τελευταίες επιβεβαιώσεις. 29 Μαρτίου το πρωί. Very Now I have four Ευχαριστώ. Έχω τέσσερις παρεμβάσεις και πρώτα το λόγο έχει η κυρία Χολ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βίκη <clears throat> για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε και γιατί ήταν τόσο κοντά στους σκιώδεις εισηγητές πράγμα το οποίο ε, είδος, ε, ίσως διαπιστώσατε με ε, τις συνενετικές τροπολογίες που θα εμπλουτίσουν το κείμενο. Πολύ χάρηκα γι' αυτό που είπες για την περιφερειακή συνεργασία για από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ανάγκη να εφαρμόσουμε καλύτερα την ισχύουσα νομοθεσία. Ε, πέραν των όσων νέων ε, θα χρειαστούν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι υπάρχει λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Δηλαδή υπάρχει συνένεση σχετικά με την σημασία του να έχει κανείς βέλτιστες πρακτικές και ασχέτως των συνθήκων να υπάρχουν οι κατάλληλες βέλτιστες πρακτικές για το χώρο αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη ε, τα οποία συμμετέχουν όντως θα εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές αλλά αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει από κοινού. Και τέλος χαίρομαι διότι αναφερθήκατε στην ανάγκη για τις εταιρείε να χρησιμοποιούν παντού τις ίδιες προδιαγραφές και εάν ε, εργάζεστε σε ένα σύστημα Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, σε ένα καθεστώς, τότε θα πρέπει ε, να γνωρίζουμε ότι ασχέτως του που δραστηριοποιείται είτε μία κοινοτική εταιρεία θα πρέπει να ε, λειτουργεί με τις ίδιες προϋποθέσεις και με την ε, ίδια αυστηρότητα να εφαρμόζει τα συμπεφωνημένα. Ευχαριστώ η κυρία Χόλη είναι ε, και ε, σκιώδης, η κυρία Καρβάλια όμως έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Βίκη ε, Φόρτ για όλα όσα μας είπε και για τον πολύ ανοιχτό και περιεκτικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται και συμπεριλαμβάνει έτσι τους συνεισηγητές. Νομίζω ότι συμφωνώ σε πολλά από όσα είπε η κυρία Φόρντ ήδη είπε ότι θα πρέπει να ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το αέριο, όχι μόνο την ε, κατάσταση του πετρελαίου, αλλά και των ε, τερματικών σταθμών ενέργειας και το αέριο κλπ. Δεύτερον, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της βιομηχανίας και των κρατών μελών. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι επαρκή πρέπει να έχουμε συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τις ε, γειτονικές χώρες. Όπως είπε και η Φιώνα Χάλ, πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό, αλλά η αεροπορική ε, η αεροπορία είναι μια βιομηχανία που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Θα έπρεπε να αναλύσουμε συνεπώς τη διαδικασία που ακολουθείται στην αεροπορία, να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποια εμπειρία από τον τομέα αυτόν, γιατί είναι δυνα... Ε, σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορούμε ε, παρά να συντονιζόμαστε σε περίπτωση που υπάρχει ένα βιομηχανικό ατύχημα. Ο ρόλος της ΕΜΣΑ επίσης ε, πρέπει να επεκταθεί, γιατί για την ώρα ο ρόλος του οργανισμού αυτού επικεντρώνεται κυρίως ε, στα πλοία, όμως μερικές φορές η εμπειρογνωμοσύνη είναι ίδια και αφορά και άλλα ζητήματα και ίσως θα έπρεπε να ε, δούμε και το θέμα της πρόληψης, της ασφάλειας και του συντονισμού ε, στον, ε, στην περίπτωση αντίδρασης σε ατύχημα ή σε κάποια κρίση στις πλατφόρμες εξόριξης αερίου ή πετρελαίου. Υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση και στο ρόλο της βιομηχανίας σε σχέση με τη βασική ευθύνη που έχει για την αντίδραση σε μια καταστροφή, για παράδειγμα. Συμφωνώ με την ιδέα ως προς τη χρηματοδότηση και την αξιοπιστία, αλλά ο συντονισμός, η πρόληψη, η ασφάλεια, η πείρα μας έχει δείξει ότι δεν είναι επαρκές, δεν επαρκής ο ρόλος της βιομηχανίας. Πρέπει ο δημόσιος τομέας ε, ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εφίσταται κάθε φορά που χρειάζεται να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μιας ε, κρίσης. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, το καταλαβαίνω γιατί οι περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές λαμβάνουν χώρα σε εκείνη την περιοχή, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, για παράδειγμα την ιδέα του φόρουμ για την ε, Βόρεια Θάλασσα και θα έπρεπε να εφαρμοστεί και στη Μεσόγειο και στον Εύξηνο Πόντο και κατά την άποψή μου οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να ζητούν ισοδύναμες προδιαγραφές. Πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν αυτό από πρακτικής απόψεως, αλλά πρέπει να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές ανεξαρτήτως του που δραστηριοποιούνται. Αυτά ήταν τα βασικά που ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σκίνερ ως ε, σκιώδης εισηγητής. Ναι, είναι γεγονό ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδου άλλο κλάδο σε σχέση με τη θνησιμότητα αν υπάρξει ε, μια καταστροφή. Εκατοντάδε ε, εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή του. Το 1988 σε αταχήματα 167 άτομα πέθαναν από τους 299 που ήταν σε μια πλατφόρμα το 1994 650 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ένα δηληστήριο στο Μεξικό και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι η προλαλή σας συνάδελφος έχει δίκιο ότι είναι σημαντικός ο ρόλος του κλάδου, αλλά πρέπει ε, να, οι προδιαγραφέ να είναι τέτοιου επίπεδου, γιατί δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια σφάλματο. Αν γίνει σφάλμα, χάνουν τη ζωή του τόσοι άνθρωποι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ επικίνδυνο εγχείρημα. Η πλατφόρμα αυτή είναι πολύ μακριά στη θάλασσα, είναι πολύ μακριά από τη στεριά για να μπορέσει να βοηθηθεί σε περίπτωση καταστροφή και, σε περίπτωση καταστροφής και είναι πολύ αργά για να γίνει οτιδήποτε. Γι' αυτό ακριβώ ο κλάδο δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε λιγότερο από τέλειες προδιαγραφές και μια σωστή και κατάλληλη ρυθμιστική προσέγγιση. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό ότι τα συνδικάτα που εκπροσωπούν τόσους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες έχουν μία άποψη για το πώς μπορούν να προστατεύσουν τους εργαζόμενούς τους και μπορεί να έχουν και ένα ρόλο ανεξάρτητο και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι σε κάθε ακρόαση θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ζητήσω από έναν ε, εκπρόσωπο των συνδικάτων. Ε, υπάρχει για παράδειγμα ε, μία, ένα συνδικάτο των Ευρωπαίων ε, εργαζομένων στη Μεσόγειο ε, στις πλατφόρμες αυτές ε, και χαίρομαι που αναφέρατε και τον αέριο, το αέριο γιατί είναι ένα ζήτημα υψηλής πίεσης ε, δεν σημαίνει βέβαια ότι το πετρέλαιο δεν, έχει, δεν αναπτύσσεται σε, υψηλό επίπεδο, σε υψηλή πίεση αλλά και το αέριο σε τέτοια πίεση δεν εξορίσεται ε, υπάρχουν τα τεχνικά επιχειρήματα, υπάρχουν οι διαδικασίες που μπορούν να μετριάσουν οποιασδήποτε συνέπειες μιας ε, καταστροφικής αδυναμίας του συστήματος. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που πρέπει να συνυπολογιστούν και γι' αυτό ακριβώς το λέω εγώ, αυτό που συμβαίνει για παράδειγμα σε βαθαία ύδατα, ε, στις για παράδειγμα, ε, πρέπει να επηρεάσει αυτό που θα κάνουμε τώρα. Πόσο χρόνο μας πήρε να εξασφαλίσουμε επιτέλους ότι θα σταματήσει η κοιλίδα. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι απαράδεκτο να πιστεύουμε ότι αν συμβεί κάποια τέτοια καταστροφή σε ευρωπαϊκά ύδατα, ότι ε, υπάρχει δυνατότητα να ανταποκριθούμε στην ε, κρίση αμέσως και πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους εποπτεία, να μην δίνουμε μόνο τη δυνατότητα στο, στους εκπροσώπους του κλάδου να μας πούν «Α, ναι, ναι, μια χαρά θα τα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε». Ε, δεν λέω ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά μπορεί να μην αρκούν οι δικέ του προσπάθειε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ω το δυνατόν τελειότερε προδιαγραφέ, όχι μόνο γιατί διακυβεύονται ανθρώπινε ζωέ, αλλά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τι ενεργειακέ μα ανάγκε. Αυτή τη στιγμή Υπάρχει μια πιθανότητα ε, ε, ε μορατόριου της πυρηνικής ενέργειας και το ίδιο μπορεί να γίνει και από το, και πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που είναι το 75% της παραγωγής μας αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια βάση μέσω της εισηγήτριας πάρα πολύ καλή για να κάνουμε πολύ διεξοδικές συζητήσεις. Ο κύριος Ρούμπιχ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Επιτροπή μας είχαμε τον εκπρόσωπο ε, της, ε, τον υπεύθυνο ασφαλείας στην Αμερική ε, και είχαμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση αλλά λόγω της καταστροφής στην Ιαπωνία πρέπει να δούμε και να κάνουμε stress test για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη θάλασσα τι θα γίνει, τι καταπονήσει υπάρχουν, αν οι τεχνικές εγκαταστάσεις είναι στο ύψος των περιστάσεων, δηλαδή θα έπρεπε να φροντίσουμε ε, δεδομένης της κατάστασης αυτής ε, να λάβουμε υπόψη την κατάσταση η οποία έχει εξελιχθεί στην Ιαπωνία. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπικ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Κατά πρώτον, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή, του συντάκτη της έκθεσης για αυτή την πρωτοβουλία. Την εισηγήτρια λοιπόν. Είναι μια χρήσιμη πρωτοβουλία, διότι έρχεται να συνεισφέρει επικοδομητικά στην όλη συζήτηση για το θέμα αυτό και βεβαίω στο έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω θα ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη σε έκθεσή τη τον Οκτώβριο αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Έγινε εκεί μια διεξοδική πολιτική ανάλυση ώστε να αναλυθεί συγκεκριμένη δράση σε τομεί που έχουν εντοπιστεί και θεωρούμε ότι η ασφάλεια των υπεράκτιων ε, εξορίξεων πρέπει να βελτιωθεί. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι η συγγήτρια και γενικώ η Επιτροπή σας, φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να συμφωνούν με τι επιτροπές που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίως ως προς τον εντοπισμό των τομέων που χρειάζεται κατευθείαν αμέσως δράση. Και του τι είδους δράση πρέπει να αναλυθεί ορισμένε φορές. Επ' αυτού, να ενημερώσω την Επιτροπή σας ότι μετά την δημοσίευση της έκθεσης τον Οκτώβριο έχουμε συνεχίσει τις εσωτερικές μας διαδικασίες απαραίτητες για την πρόθεση της έκθεσης όπως είχε προταθεί. Έγινε λοιπόν μια πρώτη μελέτη αντικτύπου η οποία εξετάζει τις ε, άμεσες συνέπειες των πρώτων δράσεων που έχουν προταθεί. Επίσης ε, πρόσφατα στις αρχές της εβδομάδας ξεκινήσαμε δημόσιες διαβουλεύσεις που θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες και θα επιτρέψουν σε όλους στην Ευρώπη να εκφράσουν την άποψή τους για το θέμα αυτό, για την υπεράκτη ασφάλεια. Και για το κοινό γιατί θα έχουμε ευρεία συμμετοχή, μιλάμε για ανοιχτά ερωτήματα. Οπότε μια μεγάλη ευκαιρία για το κοινό να εκφράσει τις απόψεις του. Όμως τα ερωτήματα επικεντρώνονται σε όλους τους τομείς που εντοπίζει η έκθεση και έχουν συνταχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρακολουθούν λίγο πολύ τη συλλογιστική της έκθεσης, της εισηγήτριά σας και τα όσα συζήτησε η Επιτροπή σας. Νομίζω λοιπόν ότι προχωρούμε, βαδίζουμε παράλληλα σε μια μορφή συνεργασίας για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε δράση θα αναλυφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θυμίζω εδώ ότι όχι μόνο η έκθεση, η ανακοίνωση μάλλον της Επιτροπής, αλλά και οι δηλώσεις του Επιτρόπου μου δείχνουν ότι η Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερος να έχει τις πρώτες πρωτοβουλίες έτοιμες ως το καλοκαίρι φέτος. Άρα δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Ιδίω με τις ολένα αυξανόμενε ανησυχίες για τον αντίκτυπο του ενεργειακού τομέα συνολικά στο περιβάλλον και την ασφάλεια παγκοσμίω. Σε αυτό λοιπόν το τοπίο, το γενικότερο τοπίο, να να πω ότι βρίσκουμε να συμβαδίζει πάρα πολύ με τις δικές μας προσπάθειες και τη συλλογιστική μας η έκθεση. Οι προκλήσεις και τα ζητήματα που θέλουμε να αντιμετωπιστούν ως τέτοια συμφωνούν και με τη δική μας οπτική γωνία. Κάποιες από τις δράσεις ή τις προτάσεις για δράσεις είναι τόσο συγκεκριμένες και χειροπιαστές και τόσο συνεπείς και με τη δική μας την ε, εξέταση του θέματος που με τα χαράς να τις εγκρίνουμε απευθείας. Ως έχουν και βεβαίω αφού εξεταστούν και μετά τη μελέτη δικτύπου και το καθεξή. Επιτρέψτε μου επίση να πω να εκφράσω μάλλον όχι επικριτικό σχόλιο, αλλά μια τρόπον την ανησυχία. Αναφέρω κάτι που και ένα από του κοιόδη εισηγητέ είπε σε μια από τι παρεμβάσει του. Αυτό που λείπει λίγο από την έκθεση που τώρα έχει υποβληθεί είναι η ευρωπαϊκή διάσταση του όλου θέματο. Υπάρχει μια σειρά από όπου δράση θα μπορούσε να αναλυφθεί. Αυτοί ορίζονται μεν, αλλά μετά η έκθεση δεν ε, διευκρινίζει ποιος πρέπει να δράσει η Ευρώπη. Θα πρέπει να δώσει όθηση στους αρμόδιους για τέτοιου είδους δράση. Θα είδατε τον Οκτώβριο στην ανακοίνωση ότι πολλές από τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν, ε, ο καλύτερος τρόπος να υλοποιηθούν είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αφήσουμε την πρωτοβουλία στα κάτι μέλη και ε, αλλά πρέπει και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν δράση. Χρειάζεται ευρωπαϊκή εμβέλεια δράση, ε, να ξεπεράσουμε τα όσα αυτή τη στιγμή αναφέρουμε ως ελάχιστα πρότυπα και να σκεφτούμε καλύτερα τις τεχνικές δυνατότητες ε, του ε, βιομηχανικού μας εξοπλισμού και τα πόσο θα κάνουμε κάποια, ή πρόβλεψη για την πρόληψη του κινδύνου. Επίσης, τι θα γίνει με τις δικαιοδοσίε και τα διασυνοριακά ζητήματα, πώ θα δοθούν οι άδειες και πώ ταυτόχρονα θα προστατεύουμε το περιβάλλον. Και το ίδιο για τις ε, βέλτιστες πρακτικές και τις ε, καλύτερες τεχνολογίες που διατίθενται. Εδώ θα υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο με ευρωπαϊκέ πολιτικέ και πρωτοβουλίε. Αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό και βεβαίω όλα αυτά μα φέρνουν στο θέμα τη διαφάνεια. Και πάλι η διαφάνεια είναι ένα παράγοντα καθοριστικό. Εκεί χρειάζεται πρωτοβουλία, ε, ανταλλαγή πληροφοριών σε όλη την Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εδώ μπορούν να αναλάβουν έναν ρόλο ζωτική σημασία. Μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο για τι πλατφόρμε για την ανταλλαγή πληροφοριών. Τέλο, η περιφερειακή συνεργασία η έκθεση καθιστά σαφές ότι εδώ οι ευρωπαϊκοί φορείς μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Νομίζω λοιπόν χρήσιμο θα ήταν να σκεφτούμε και άλλα ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται αναγκαστικά στην έκθεση όταν σκεφτόμαστε στην ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος. Ευχαριστούμε κυρία Φόρτ. Η κυρία Φόρτ και πάλι αλλά σύντομα γιατί έχουμε μισή ώρα για το επόμενο θέμα. Άρα μισό λεπτό τώρα. Λοιπόν, συμφωνώ σχεδόν πλήρως με όσα ελέγχθησαν. Προφανώς ε, υπάρχει μία θέση για την ΕΜΣΑ σε ε, περίπτωση μίας καταστροφής θα ήθελα η ΕΜΣΑ να εξασφαλίσει ότι οι χώρες θα μιλούν με μία φωνή και με μία ε, κοινή ορολογία για να συντονίζονται σε περίπτωση καταστροφής και όταν λέγω ότι είναι πρώτη ευθύνη εννοώ για να υπάρξουν εγκαίρως οι και να έχουν καταβληθεί εκ προημίου σε περίπτωση μίας καταστροφής. Αυτό λέγω ότι είναι κάτι που θα πρέπει οι αρχές να σκεφτούν για να είμαστε δίκοι ότι θα υπάρχει συντονισμός όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις γειτονικές χώρες για τις καλές πρακτικές ε, αδειοδοτήσεως συμφωνώ μαζί σας για την διαφάνεια της βιομηχανίας και τον καταμερισμό των βελτίστων πρακτικών βεβαίως θα πρέπει να επικοινωνούμε περισσότερο διεθνώς και όχι μόνο εντός της Ευρώπης των 27 ε, το πρότυπο των αεροπορικών εταιριών παραδείγματο χάρη είναι πανευρωπαϊκό και όχι μόνο είναι, παγκόσμιο και όχι μόνο πανευρωπαϊκό. Επίσης ε, όσον αφορά το, τα θέματα περιβάλλοντος χαιρετίζω την επιθυμία των μελών της Αρμόδιας Επιτροπής να συμμετάσχουν, να μου κάνουν ένα τηλέφωνο και ευχαρίστως θα συνεργαστούμε. Ε, ε, τώρα το θέμα των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη θάλασσα, offshore, και σε σχέση ε, με αυτές που βρίσκονται στην ξηρά. Είχαμε προσφα... προετών στην περιοχή μου μία φοβερή καταστροφή σε ένα δηληστήριο και όντως πρέπει να υπάρχει συντονισμός. Όσον αφορά τη γύραση των εγκαταστάσεων, σας ευχαριστώ και κοιτάζω τα συμπεράσματα της Ιαπωνίας ε, θα πρέπει να το επανεξετάσουμε σε πέντε χρόνια διότι αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει και πριν από λίγα χρόνια ε, έκτοτε νομίζω ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει και μπορούμε τώρα να δούμε ε, εάν ε, όντως υπάρχουν ευέλτιστες πρακτικές για να διεκπαιρεώσει κανείς τα θέματα αυτά. Διότι ε, πρέπει ε, να υπάρξει μια κατάσταση η οποία να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν και σύμφωνο ότι πρέπει να είναι ασφαλής. Αυτά. Αυτά είχα να σας πω, πολλά πρέπει να κάνουμε, αλλά αυτά είχα να σχολιάσω τώρα. Ωραία, και τώρα ένα λεπτό. Όχι, δεν έχουμε προθεσμίες, οπότε τώρα μιλάμε για την ακεραιότητα και διαφάνεια της αγοράς ενεργείας. Ο κύριος Χατζημαρκάκης για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα μιλάμε για την ακεραιότητα και διαφάνεια της αγοράς ενεργείας. Είναι μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ρύθμιση του τομέα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των χρηματοοικονομικών αγορών. Και ε, σήμερα έχουμε τον κύριο Γκέμπελς εδώ, ο οποίος είναι και μέρος της αρμόδιας επιτροπής και ε, ασχολείται με χρόνια στα, με τα θέματα της ε, κακής διαχείρισης των ε, χρηματαγορών και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά νέα μέσα, φιντ και ούτω καθεξής αλλά στον τομέα των παραγωγών και των εμπόρων ενεργειών θα χρειαστούμε μία συγκεκριμένη ε, νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν μία πρόταση η οποία ε, επανέρχεται στα θέματα που είχε θίξει και ο Ρόμπερτ Γκέμπερ στο 2003 είναι προσαρμοσμένο στις χρηματοοικονομικές δομές ή στον ενεργειακό τομέα. Γιατί τις χρειαζόμαστε. Διότι μέσω των ε, χρηματοοικονομικών παραγόγων οι τιμές της ενεργείας εξασφαλίζονται μακροπρόθεσμα αλλά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, τους εμπόρους ενέργειας όπως τις τράπεζες και σχετικά με τη MIFID παραδείγματος χάρη θα πρέπει να μην, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι έμποροι ενεργείες για τεράστια ποσά όπως οι τράπεζες. Αλλά όταν μιλάμε και για ανοιχτές συναλλαγές ε, μεταξύ εμπόρων τηλεφωνικά και γενικότερα ε, υπάρχει ένας τεράστιος τομέας όπου μπορούν να υπάρξουν παρεκτροπές. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε με την πρόταση αυτή ε, οδηγίας είναι να έχουμε ένα σύστημα ανακοίνωσης για το πετρέλαιο και το αέριο κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσει να λειτουργήσει η επιτροπή που δημιουργήθηκε την περασμένη εβδομάδα η Acer η οποία έχει έδρα στην Λουμπλιάνα και ε, όπου συμμετέχουν οι ρυθμιστίες του τομέα μας για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν στοιχεία από τις ε, πράξεις οι οποίες γίνονται εκτός χρηματιστηρίου. Ως εδώ πάμε καλά. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα κράτη όπως αυτό του Προέδρου το οποίο, τον οποίο γνωρίζω πολύ καλά, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν στη χώρα μία άλλη οργάνωση για τη διαφάνεια της αγοράς. Εάν όμως θέλουμε να πάμε μπροστά πρέπει να υπάρχει μία ευρωπαϊκή αρχή που να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και για το αέριο και για τον ηλεκτρισμό και ε, για το διοξίδιο του άνθρακος όπου υπάρχουν τα πιστοποιητικά και το εμπόριο διοξιδίου του άνθρακος και ε, ε, δεν μπορούμε να αποδεσμεύσουμε το διοξίδιο του άνθρακος από τον ηλεκτρισμό και το αέριο και γι' αυτό κάνω μία έκκληση να ασχοληθούμε και με το διοξίδιο του άνθρακος διότι διαφορετικά δεν υπάρχει κανένα νόημα. Όσον αφορά τον άνθρακα και το πετρέλαιο ε, υπάρχει μία σφαιρική αντιμετώπιση αλλά δεν μπορούμε εδώ να παραβλέψουμε το διοξίδιο του άνθρακος δεν βλέπω γιατί πρέπει να το αποδεσμεύσουμε και να το ξεχωρίσουμε επειδή έχουμε ε, δύο διαφορετικούς ε, επιτρόπους ε, τον κύριο Έτιγκερ και τον υπεύθυνο για το περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει στην ανακοίνηση αυτή να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει τα στοιχεία ε, να πηγαίνουν ε, ή στην ε, ΑΣΕΡ στον αρμόδιο οργανισμό και να είναι μονόδρομος αυτή η διαδικασία και στη συνέχεια να εμπλέκονται τα κράτη. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει αυτό να περιληφθεί στην νομοθεσία αυτή, ότι η Acer θα είναι η ρυθμιστική αρχή η οποία θα ενημερώνεται όποτε υπάρχει στρέβλωση της διαχειρήσεως της αγοράς. Ένας συνομιλητής πρέπει να υπάρχει για ρυθμιστικούς στόχους και μετά θα υπάρξουν αρχές οι οποίες ασχολούνται με ε, την διαφθορά και τη στρέβλωση και θα επεμβαίνουν αλλά ο ρυθμιστής πρέπει να είναι ο πρώτος συνομιλιστής μας. Αν όλα γινόντουσαν μέσω χρηματιστηρίου, όλες δηλαδή οι πράξεις διεξαγόντουσαν μέσω χρηματιστηρίου, θα μπορούσαμε να, πά, να τα ελέγξουμε καλύτερα, αλλά 60 μέχρι 80% των πράξεων διεξάγονται εκτός χρηματιστηρίου. Όταν λοιπόν μιλάμε ε, ε, για εκμετάλλευση της αγοράς, θα πρέπει να έχουμε μία ενιαία εναρμονισμένη διαδικασία διότι τι θα γίνει διαφορετικά αν υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής τότε το εμπόριο το οποίο που παρακάμπτει την ομοθεσία θα αναπτυχθεί και γι' αυτό χρειαζόμαστε και κυρώσεις εναρμονισμένες. Τι θα γίνει με το επίπεδο των κυρώσεων. Εδώ είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να σκεφτούμε ε, τουλάχιστον περιθώρια de ελάχιστα, τα οποία όμως δεν πρόκειται εμείς να ρυθμίσουμε τώρα. Θα είναι μία εντεταλμένη πράξη που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα πρέπει τα delegated acts να περιοριστούν σε συγκεκριμένους στόχους για να δούμε πότε θα ισχύει ο κανόνας de minimis και πότε θα χρειαστεί να εμπλακεί ένα delegated act το οποίο θα αναλάβει να ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό ο αδειοδοτήσεως. Υπάρχει ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο τα κράτη ε, ε, ε, προβαίνουν εις τις αιτήσει, αλλά χρειαζόμαστε ένα κοινοτικό σύστημα για την αδειοδότηση. Δεν χρειάζεται εδώ να έχουν εγγραφεί όλοι οι μικροέμποροι, αλλά τουλάχιστον οι μεγαλέμποροι χρειάζεται να έχουν έχουν καταγραφεί για να μπορούμε να ελέγξουμε την πρόταση. Ε, διότι βλέπουμε ότι σε άλλα κράτη υπάρχουν οργανώσεις όπως η Άσερ και ε, εκεί υπάρχουν και περισσότεροι υπάλληλοι από τους 25 που προβλέπουμε εδώ. Πιστεύω ότι 25 είναι λίγοι διότι για να παρακολουθεί κανείς τη ροή των δεδομένων χρειαζόμαστε περισσότερα άτομα και χρειαζόμαστε και ένα ή δύο ε, ε, γραφείο σύνδεσμο. Δεν ε, μπορώ να σκεφτώ πού θα ιδρεύσει, ίσως στην Ευρωπαϊ... στις Βρυξέλλες για να είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορέσει να συνδυαστεί με τον χώρο που συγκεντρώνονται και συνεδριάζουν οι εθνικοί ρυθμιστές αλλά όταν έχετε γραφεία συνδέσμων είσαστε πιο κοντά στην αγορά ίσως και το Λουξεμβούργο θα ήταν μία λύση η Λουμπιάνα είναι εξαιρετική αλλά ε, υπάρχουν προβλήματα με τα παιδιά διότι τα υψηλά στελέχη έχουν οικογένειες και Τέλος, ουσιαστικό θέμα είναι οι ορισμοί, οι οποίοι ε, είναι ξεπατήκωμα του ότι είχε ε, χρησιμοποιήσει ο κύριος Γκέμπελς προετών και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι. Πρέπει να διαφοροποιούμε μεταξύ της αγοράς ηλεκτρισμού και αγοράς αερίου διότι υπάρχουν διαφορετικοί μηχανισμοί τους οποίους πρέπει να διευκρινίσουμε ε, πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ ε, της ε, ανακοινώσεως των ατόμων ή της ανακοινώσεως των πράξεων και πρέπει να κλείσουμε τα κενά προς την ΜΥΦΙΤ ε, και άλλες οδηγίες. Θα πρέπει να υπάρξει μια στενότερη ε, σχέση μεταξύ της ε, Άσερ και της ΕΣΜΑ την οποία αποφασίσαμε πριν λίγο καιρό και γι' αυτό θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον ο κύριο Γκέμπελς και τον κύριο Σβόμποντα με τους οποίους θα ξανασυναντηθώ για την εξαιρετική συνεργασία μέχρι τώρα. Ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουν να ακολουθήσουν και οι συνάδελφοι τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ, ο κύριος Σουάμποντα. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Αυτό που είναι ουσιαστικό είναι να έχουμε αλλαγή στον τομέα αυτό ε, και γι' αυτό νομίζω ότι καλό θα ήταν να περιληφθεί και το θέμα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Ορισμένοι θέλουν να υπάρχει σοβαρή ε, ρύθμιση και αυτό βέβαια το προτιμούν οι σοβαρές ε, εταιρείε και θα πρέπει να έχουμε ένα καλό σύστημα πληροφόρησης διαφορετικά θα υπάρχει σύγχυση συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Χατζημαρχάκης για τον ορισμό. Δεν μπορεί αυτό να αναλυφθεί από τα Delegated Acts, διότι αν πρέπει από τόμος ε, να κλείσει μία μονάδα ένας παραγωγός ενεργείας, και ε, εάν αυτή η μονάδα ασχολείται με την παραγωγή ηλεκτρισμού τι θα γίνει, είναι της δικαιοδοσίας του ή όχι. Ε, το θέμα δεν είναι να επιβάλλουμε κυρώσεις αλλά να υπάρχει λογική αντιμετώπιση. Και τέλος ε, πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει σχετικά με τις εθνικές αρχές και τις ποινές διότι δεν σημαίνει ότι οι χώρες οι οποίες ε, ε, ε, δεν εφαρμόζουν τα συμπεφωνημένα να έχουν περισσότερη δουλειά διότι μπορούν να παρακάμψουν τις κυρώσεις. Ο κύριος Γκέρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν Ευχαριστώ. Υπάρχει μια ενεργειακή πολιτική η οποία δεν χρειάζεται νέες πολιτικές αλλά εφαρμογή των ισχυουσών πολιτικών, βελτίωση των υποδομών και μετά νέες ρυθμίσεις διότι ε, η περίπτωση που εξετάζουμε είναι μια εξαίρεση ε, διότι χρειάζεται διαφάνεια των αγορών και αυτό πρέπει να επιτευχθεί παράλληλα προς τις παλαιότερες διαδικασίες δηλαδή στη βελτίωση των υποδομών και γι' αυτό χρειάζεται μια ευρωπαϊκή νομοθεσία διότι δεν μπορεί να καλυφθεί το θέμα από τις εθνικές νομοθεσίες εξού και ε, πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το ε, πρόγραμμα των τραπεζών. Ε, πιστεύω δε ότι ο τομέας αυτός θα μπορέσει να μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μία συνένεση σε έναν τομέα ο οποίος πλήττεται από την κρίση και να επιτύχουμε τη συνένεση αυτή σε πρώτη ανάγνωση. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα το οποίο έθεσε και ο εισηγητής ε, και θέλω να τονίσω εγώ και άλλα τέσσερα θέματα. Καταρχήν, θα σε ποιον θα απευθύνονται οι έμποροι για να αποδώσουν τα στοιχεία τους. Δεύτερον, πώς θα συγκεντρώνουν τα στοιχεία, πώς θα προστατεύονται και τέταρτον, κυρώσεις. Και προσπαθώ να είμαι πολύ σύντομος. Πρώτο ερώτημα, ποιος θα συγκεντρώνει τα στοιχεία. Ξέρω ότι το Συμβούλιο ε, δεν ε, συμφωνεί ε, στο θέμα αυτό, είναι διηρεμένο και πρέπει να προχωρήσουμε διότι καταρχήν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μέσω του κεντρικού οργανισμού και μεταξύ των γραφείων εποπτείας θα μπορούν να συγκεντρώνουν περισσότερα στοιχεία που θα προέρχονται από την αγορά. Άρα λογικά ε, θα έπρεπε ο οργανισμός που είναι στη Λουμπλιάνα να χρησιμοποιηθεί σαν συντονιστικό σημείο. Ξέρουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει το καλύτερο ευρωπαϊκό σχολείο στην Λουμπλιάνα, δεν ε, ξέρω ποιο είναι το καλύτερο σημείο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να εδρεύσει η εταιρεία αυτή, αλλά είναι κάτι το οποίο ίσως μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια. Δεύτερον, όσον αφορά τον τρόπο της ε, παραδόσεως των στοιχείων, δηλαδή ε, πώς θα μεταδίδονται τα στοιχεία ή στο γραφείο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει επιλέξει τη διαδικασία του Delegated Act και δεν διαφωνούμε διότι θα πρέπει να ε, μπορούμε να προχωρήσουμε και μέσω αυτής της μεθόδου αλλά πρέπει σαφώς αυτά τα στοιχεία να είναι λεπτομερή θα πρέπει ε, να ε, ακολουθήσουν την, το πνεύμα της ε, συγκεντρώσεώς τους ε, για να μπορέσουν ε, να συνεκτιμηθούν σωστά και να δούμε πώς θα τα πλαισιώσουμε. Και τέλος όσο αναφορά την προστασία των στοιχείων πρέπει να πούμε ότι είναι ευαίσθητα στοιχεία τα οποία μεταβιβάζονται και αν προωθηθούν και εις τους ανταγωνιστές εκτός γραφείου τότε αυτά τα στοιχεία θα μπορούν ε, να διανεμηθούν πέραν του κύκλου που επιθυμούμε ε, και πρέπει να βρούμε τρόπο να τα προστατεύσουμε. Τέλος, ε, κυρώσεις. Αντιλαμβάνουμε την ανησυχία ότι θα πρέπει να υπάρξουν διαφορετικές κυρώσεις και ε, να ε, ε, μην ε, μπορούν οι έμποροι να παραμείνουν στα κράτη όπου υπάρχουν λιγότερες κυρώσεις αλλά υπάρχουν εδώ και αρμοδιότητες των κρατών και θα πρέπει να βρούμε μία συμβιβαστική πρόταση. Ευχαριστώ και ελπίζω θα έχουμε χρόνο για περαιτέρω σχόλια. Τέλος θα ήθελα να πω ότι εάν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε, αυτή τη, σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πρώτη ανάγνωση. Και τώρα έχουμε 8 λεπτά για του υπόλοιπου ομιλητέ εκ των οποίων ο πρώτο ο κύριο Γκέμπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ταχύτατα. Είμαι εισηγητή για την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και έχω αποβάλει τη δικά μας σχόλια στην γραμματεία της Επιτροπής. Θα θέλαμε και η δική σας λοιπόν επιτροπή να ετοιμάσει τη γνωμοδότησή όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε τα στοιχεία μας τα στοιχεία μας να μπορέσουν να αξιοποιηθούν από τον κύριο Χατζημαρκάκη, στον οποίο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Πρώτη παρατήρηση. Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν και αγορές ε, OTC, γιατί εκεί υπάρχουν άμεσες συμβάσεις που δεν παίρνουν από τι ρυθμισμένε αγορές. Μιλήσατε επίσης για την ανάγκη να πρικοδοτήσουμε με πόρους τους φορείς, ναι, διότι αν δεν τα έχουμε τα απαραίτητα μέσα, δεν θα αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος. Και παραμένει το πρόβλημα των ερισμών. Όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπνεύστηκε από την οδηγία για την κατάχρηση στις αγορές, αλλά και από την συζήτηση του Κοινοβουλίου που είχε γίνει όταν ξεκίνησε η συζήτηση για εκείνη την οδηγία. Διότι αν τελικά η πρόταση. και όμω θα έχουμε προβλήματα συνέπειε ακριβώ γιατί αν η τωρινή οδηγία έγκριθει ή απορριφθεί, θα επηρεαστεί αναλόγω και η προηγούμενη για την κατάχρηση των αγορών. Εδώ χρειάζονται εξελαχίστων κανόνε ούτω ή άλλω. Διότι θα συγκεντρώσουμε ένα πλήθο περιττών πληροφοριών και οι μεγάλε συναλλαγέ πρέπει να περιορίζονται από κάποιο ανώτατο όριο. Και αυτό θα γίνει μόνο από δευτερογενή πράξη, πράξη κατά εξουσιοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να ρίξει και εκεί μια ματιά. Έπειτα ένα σύστημα κυρώσεων αποτελεσματικό. Ο συνάδελφος δίκιο έχει, που λέει ότι αν δεν προβλεφθεί αυτό, euh, μπορεί να έχουμε εμπορευόμενου που θα καταλήγουν να εγκαθίστανται στι χώρε όπου υπάρχουν λιγότερε κυρώσεις. Αυτό δεν πρέπει να επιτρέπεται. Θα πρέπει να, υπάρχει ισότιμη, ισότιμη, να υπάρχουν ισότιμοι κανόνε για όλου του εμπλοκόμενου και να του ρυθμίζουν οι εθνικοί νομοθέτε και ρυθμιστέ. Θα πρέπει να υπάρχουν όμω και σε ευρωπαϊκό σύστημα κάποιε προβλέψει ώστε οι κυρώσει να είναι αποτελεσματικέ και ανάλογε με τα ενδεχόμενα κέρδη ή απώλειες. Τελευταία παρατήρηση Ο φίλος ε, κ. Χατζημαρκάκης συμπεριλαμβάνει και τις αγορές για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. δεν έχω αντιρρήσει προς την πρότασή του, διότι είδαμε ότι στην αγορά του διοξιδίου υπήρξαν ατασταλίες και κάποιες παρανομίες που ανακαλύφθηκαν, σίγουρα κάποια πέρασαν απαρατήρητα, αλλά υπήρξαν και απάτες και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ε, κατά κάποιων χρηματιστηρίων για αυτές τις περιπτώσεις εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Να τα σκεφτούμε λοιπόν όλα αυτά προσεκτικά. Η κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ακριβώς αυτό που μόλις είπε ο κύριος Γκέμπελς. σε σχέση με την αγορά αδειών εκπομπών. Υπήρξαν πολλές απάτες ε, και μέσω της τεχνολογίας των υπολογιστών και πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε το μάθημά μας. Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει πλήρης διαφάνεια της ε, αγοράς ενέργειας. Και το λέω αυτό γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυξάνονται οι τιμές, έχουμε όλο και περισσότερο δυσκολία ε, ο κόσμος να πληρώνει τους ενεργειακούς του λογαριασμούς και θα πέσει κάτω από το αποδεκτό, από το κατόφλι της φτώχειας. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς. Επομένως, καλό θα ήταν όλοι να καταλαβούν πώς υπολογίζεται μία τιμή της ενέργειας. Όσον αφορά τώρα ο φόρο, το, το φόρο προστιθέμενης αξίας που είναι διαφορετικός από τη μία χώρα στην άλλη και από το ένα προϊόν στο άλλο, στο τομέα της ενέργειας τουλάχιστον νομίζω ότι ο ΦΠΑ έχει επίσης πάρα πολύ σημαντική επιρροή στην τελική τιμή που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής. Ο κύριος Ρούμπικ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο παρατηρήσεις. Στην Αμερική ε, κατάφεραν να διαφορήσουν τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές από το φυσικό εμπόριο του προϊόντος. Οπότε αυτό θα έπρεπε να πετύχουμε και εμείς και όσον αφορά τις εκπομπές διεξιδίου του άνθρακος όντως πρέπει να αποδεικνύουμε ποιες είναι οι ουσιαστικές ποσότητες που πουλάμε και ποιες είναι οι ιδεατές, οι χρηματιστηριακές. Βέβαια όταν τελειώσει αυτή η κρίση στην Ιαπωνία θα πρέπει να αποκομίσουμε ε, τα συμπεράσματα και να δούμε τι σημαίνει αυτή η κρίση για την Ευρώπη. Θα είναι ε, πιο δύσκολο για να επιτύχουμε αυτή τη μείωση και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι στόχοι μας θα χρειαστεί ίσως ε, να υποβιβαστούν διότι ε, το ποσοστό αυτό που είναι ελάχιστο της χιλής ε, μας δίνει μία ικανοποιητική ε, απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα με σύντομο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Χαίρομαι όλο ιδιαίτερο που ο κύριο Χατζημαρκάκη ε, αντιμετώπισε ένα τέτοιο πολύ περίπλοκο ζήτημα τόσο καλά είπε ότι είναι εντελώ ετερογενής η κατάσταση και ότι είναι διαφορετική η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Οπότε πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγουμε κάποιους κανόνες. Χρειάζεται να έχουμε ενιαίους κανόνες για τους εθνικούς ρυθμιστές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η διαθέσιμη πληροφόρηση είναι ε, συγκρίσιμη, ότι τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα. Και είναι σημαντικό να έχουμε και πολύ σαφείς κανόνες σε σχέση με τις ε, πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες. Νομίζω ότι αυτό λοιπόν είναι εξαιρετική σημασία ζήτημα. Και μάλιστα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν σαφώς καθορισμένους κανόνες και να συνεχίσει η συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και υπάρχουν και με διαφορές σε σχέση με τις ανησυχίες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη για την ε, ε, κατάχρηση των δεδομένων, για την κακή χρήση των δεδομένων. Είναι επίσης και διαφορετικό το επίπεδο της διαφθοράς σε κάθε κράτος μέλος και η πίεση είναι τεράστια. Και εγώ ευχαρίστως να συνεργαστώ με τον κύριο Χατζημαρκάκη και χαίρομαι ιδιαίτερα που συζητούμε το θέμα αυτό σήμερα. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή πρέπει να παρέμβει. Παρακαλώ όμως να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ για την ε, δυνατότητα. Και ευχαριστούμε που εξετάζετε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα με τέτοιο ενθουσιασμό. Τα ζητήματα που προέκυψαν στην συζήτηση μας καταδεικνύουν τη σωστή κατεύθυνση. Έχετε καταλάβει ορθώς το θέμα. Um, ήδη <laughs> είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τις απόψεις των μελών εδώ στην αίθουσα και ακούσαμε και έχουμε καταγράψει ήδη τις παρατηρήσεις τους. Πολλές έχουν ήδη ακουστεί και σε συζητήσεις του Συμβουλίου στην ομάδα εργασίας της ενέργειας. Είμαστε λοιπόν ήσυχοι ότι τα θέματα που θέσατε με τον ένα τον άλλο τρόπο θα λυθούν. Κάποια μάλιστα είχαν εξεταστεί λεπτομερώς. Όποια βοήθεια χρειαστείτε, όποια διμερή συνάντηση, με μεγάλη μας χαρά να σας τη δώσουμε. Για όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν. Ευχαριστώ. Και τέλος ο συνάδελφος Χατζηματικάκης Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία και για τη συνένεση, ιδίως σε θέματα τόσο λεπτά όσο η εμπορία του διοξιδίου του άνθρακος. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είχαμε εξαιρετικές συναντήσεις όπου παρίσταντο διάφοροι συνάδελφοι και πιστεύω ότι μπορούμε να το κλείσουμε σε πρώτη ανάγνωση ε, στο δεύτερο εξάμεινο ή στην ε, ε, Πολωνική Προεδρία έχουμε πολλούς φακέλους έχουμε και το REMIT το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και αυτό τα προβλήματα είναι τεχνικά αλλά πιστεύω ότι ουσιαστικά θα έχουμε προχωρήσει εγώ θα έχω ολοκληρώσει την έκθεσή μου την επόμενη εβδομάδα, άντε το πολύ την ε, μεθεπόμενη και ε, τον τέλη Απριλίου θα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες κατά τρόπον ώστε η Ρέμιτ να ε, ψηφιστεί στην Επιτροπή τέλος Μαΐου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ιδίως για την ταχύτητα και ευχαριστώ και τους διερμηνείς οι οποίοι μας βοήθησαν να μείνουμε λίγα λεπτά παραπάνω και σας υπενθυμίζω αύριο την ε, ε, ακρόαση για τις ε, διαρροές διοξιδίου του άνθρακος και για την εμπορία των, των εκπομπών και σας εύχομαι καλή μέρα.